Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δημογραφική αλλαγή και η ισορροπία, η δίκαιη αντιμετώπιση των γενναίων είναι το θέμα μου. Βασίζομαι σε μία σειρά από μελέτες που έχουν γίνει σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ήρθα σε επαφή με πολλούς φορείς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτός και είχα και την ευκαιρία να μιλήσω με ΜΚΟ και με προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάναμε επίσης και ένα μικρό hearing εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η κατά κάποιο τρόπο θέση κίνησής μας. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι γυράσκουν όλο και περισσότερο, ζουν περισσότερα χρόνια, ζουν με υγεία όλο και περισσότερα χρόνια. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή ότι μπορούν να παραμείνουν ενεργοί πολύ περισσότερο. Δεν νομίζω λοιπόν δυνατικό ότι υπάρχει αυτή η γύρανση, η ενεργή γύρανση. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικούς, με δημοσιονομικούς κινδύνους ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των καθεστώτων συντάξεων. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε εγκαίρως και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό το οποίο έγινε σε ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ουσιαστικά έχει τεθεί αντιμέτωπη μία γενιά εναντίον των άλλων και τσακώνονται διότι λέει ο ένας τα δικά μου συμφέροντα πιο σημαντικά από τα άλλα. Επομένως, για μένα πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή ωφελών και υποχρεώσεων μεταξύ των γενεών. Αυτό σημαίνει για μένα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φυσικά θα λάβει υπόψη και τι εμπειρίε των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε ένα ανοιχτό διάλογο μεταξύ των γενεών και θα πρέπει να αποφύγουμε τις πολεμικές και αντιπαραθετικές αντιμετώπισης για να έχουμε μια λύση που θα είναι win-win, θα είναι θετικού αθροίσματος για όλους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε τα εργαλεία πληροφόρηση, να έχουμε ένα φόρουμ σε κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία να βλέπουμε πώ θα εξελίσσεται η κατάσταση στο μέλλον. Τι πληρωμέ απαιτούνται, τι επιβαρύνσει θα προκύψουν από την αλλαγή τη δημογραφική ισορροπία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μία <clears throat> αξιολόγηση τη κατάσταση αυτή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι γνώσεις μας να μην μένουν στα αρχεία, αλλά να χρησιμοποιούνται ενεργά και να μπορούμε να δούμε ποια ακριβώς είναι η επίπτωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, να γίνουν επομένω ορατά όλα αυτά. Όλα αυτά απαιτούν πλατφόρμες επικοινωνίας μεταξύ των γενναίων. Αυτό δεν αφορά λοιπόν μοναχα του νέου και του ηλικιωμένου. Όλη τη την κοινωνία μα πρέπει να εμπλέξουμε ώστε να έχουν όλη την ευθύνη για τι μελλοντικέ εξελίξει. Επομένω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπέρχει και μια εγγύηση σε σχέση για του νέου, η ενεργία των νέων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που οδηγεί σε μεγάλο εξοπλισμό και φυσικά και σε μια τεράστια σπατάλη ανθρωπίνων πόρων και δεξιοτήτων. Και βλέπουμε ότι οι νέοι ότι αντί να <clears throat> συμμετέχουν στην κοινωνία, αντί να είναι τμήματα της κοινωνίας, έχουν μια στάση απόρριψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί θα πρέπει μετά από ανεργία έξι μηνών το μέγιστο, ο κάθε νέος να έχει τη δυνατότητα μιας θέσης μαθητείας ή κατάρτισης για να μπορέσει να συνεχίσει την εργασιακή του καριέρα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταβάλουμε τις προσπάθειες αυτές για να εξασφαλίσουμε και την ενσωμάτωση των νέων στην κοινωνία. Όχι λοιπόν να, και από την πλευρά των νέων όχι μόνο να περιμένουν παθητικά την υποστήριξη από το κράτος, αλλά να είναι και αυτοί ενεργοί στην αναζήτηση λύσεων. Να μην μείνουν λοιπόν εκτός της αγοράς εργασίας για πολύ καιρό οι νέοι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτά αφορούσαν τους νέους. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους χρειάζεται μια νέα συν... κατά κάποιο τρόπο μια νέα σύμβαση με τους ηλικιωμένους που είναι πάνω από 50 ετών. Δεν θα πρέπει αυτοί να αποκλείονται από την αγορά εργασία, να υποχρεώνται να εγκαταλείψουν την ε, <clears throat> αγορά εργασία, αλλά πρέπει να νιώθουν ότι του χρειάζονται, ότι είναι αγαπητοί στην αγορά εργασία, ότι υπάρχει δυνατότητα να συνεργάζονται με του νέου σε κοινέ ομάδε εργασία, κάτι το οποίο οδηγεί σε αμοιβαία ωφέλη και για τους νέους οι οποίοι μπορούν να επωφελούνται από την πείρα των ηλικιωμένων και από τους ηλικιωμένους οι οποίοι μπορούν να ωφελούνται από τις νέες ιδέες των νέων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ως πολιτικοί να πείσουμε τις επιχειρήσεις, τους μάνατζερ, τους κοινωνικούς εταίρους, τα συνδικάτα να παίξουν το ρόλο τους μέσα σε αυτόν τον χώρο και να γίνουν οι απαραίτητες ε, αλλαγές. Χρειαζόμαστε να δώσουμε κίνητρα στους ηλικιωμένους άνω των 60 για να παραμείνουν στη θέση εργασία τους, εφόσον φυσικά είναι σε επαρκή κατάσταση υγείας. Αυτό συμβαίνει πια. Υπάρχουν λεγόμενοι νέοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τη δυναμικότητα που είχαν παλιά οι άνθρωποι 40 ετών. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να είναι μια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ικανοτήτων και των προσφορών που μπορούν να αναδώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Χρειάζεται μια πρωτοβουλία, όπως την είπα, age management, δηλαδή μια διαδικασία η οποία προωθεί την ενεργό γύρανση, και μια σειρά πρωτοβουλίων προς την κατεύθυνση αυτή και βασίζομαι και στην συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των συνδικάτων που είναι απαραίτητη για τον τομέα αυτό. Έχω προτείνει επίσης στον τομέα της ε, οικονομικής ανάπτυξης ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα την οικονομία που περιστρέφεται γύρω από τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, πολλές υπηρεσίες που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά αυτό δεν φτάνει. Μπορεί να λέει ένας νέος ότι αυτό είναι μονάχα για τους γέρους. Ή μπορεί να πει κάποιος ότι λόγω αυτής της ενασχόλησης μόνο με τους νέους στην αγορά, στα μέσα ενημέρωσης και στα κόμματα, οι γέροι δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό είναι μια αρνητική αντιμετώπιση, μια αρνητική κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί και πρέπει να την αποφύγουμε. Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το θέμα της περίθαλψης των ηλικιωμένων. Έχουμε διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων φεύγει από τις περιοχές της υπαίθρου, δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί. βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν είναι παρόντες οι ηλικιωμένοι για, σε, σε τέτοιες περιοχές υπαίθρου. Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε επομένως τις ε, πρωτοβουλίες αυτές, ώστε στις περιοχές αυτές οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα όταν βρουν μια θέση κατάρτιση, μια θέση εργασίας να έχουν, να και από την εμπειρία των πιο ηλικιωμένων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Ένα τμήμα της Γερμανίας έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αν οι πολιτικοί θέλουν να έχουν κάποια επιρροή στη λειτουργία της κοινωνίας θα πρέπει να επηρεάσουν και τη σχέση των νέων με τους ηλικιωμένους. Ε, στον τομέα της περίθαλψης συγκεκριμένα είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, όχι να λένε ότι μπορούμε κάπου να αφήσουμε τους ηλικιωμένους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες κάπου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συμμετοχή όλων σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως ε, μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ε, πρόκειται ε, για το εξής πρόβλημα. Ε, μερικές φορές τους λείπουν και τα κατάλληλα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή, αλλά και τα χρήματα. Για σκεφτείτε, στις δημόσιες υπηρεσίες οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία και από τους παλιούς και να δουν τι ακριβώς γινόταν. Και εγώ είδα με τι επαφές μου ότι οι νέοι πολλές φορές υποστηρίζουν ότι ε, οι ηλικιωμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν και να ε, χειρίζονται το ίντερνετ καλύτερα από τους νέους. Άρα λοιπόν το θέμα είναι θέμα πρόσβασης. Αν έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι τέτοιο, αν έχουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτές τις εξελίξεις. Και αυτές οι ενεργές παροχές που μπορούν να προκύψουν από τους ε, ηλικιωμένου δεν είναι να διδάσκουν από καθέδρας, αλλά πρώτα να δίνουν την εμπειρία Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή επομένω προσπαθεί όχι να δει τα πράγματα μονάχα από την πλευρά των ηλικιωμένων ή από την πλευρά των νέων, αλλά να συνδυάσει και να συμβιβάσει τις δύο απόψεις. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε μεταξύ των δύο πλευρών. Ξέρουμε ότι το σύστημά μας Τη κοινωνική ασφάλειας κάποια στιγμή θα καταλήξει στο από τη ιστορίας εάν δεν επιβάλλουμε κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσει σε αυτό το σύστημα. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια κοινή πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να συζητήσω τα θέματα αυτά μαζί σα. Thank ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στην ε, πρώτη ομιλητρία, στην κυρία Κουνέλσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, Πρέπει ε, Κορνέλισεν, συγγνώμη, χαίρομαι πολύ για το γεγονό ότι έχουμε αυτή την έκθεση και οι δημογραφικέ αλλαγέ πραγματικά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή συζητάμε ε, ιδιαίτερα ε, για την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν σήμερα χώρε τη Ευρώπη. Πιστεύω όμω, ότι η βιωσιμότητα ε, του, των ε, συνταξιβετικών συστημάτων κυρίω και η δημογραφική αλλαγή είναι κάτι το οποίο μα περιμένει στη γωνία και η κρίση θα ξεσπάσει αν δεν κάνουμε κάτι. Ταυτόχρονα συμφωνώ με τον κύριο Μαν ε, για το γεγονό ότι είμαι πεπισμένη ότι η δημογραφική αλλαγή ε, είναι διαχειρίσιμη, αν όμω ε, την προβλέψουμε στον σωστό βαθμό. Και εδώ η έκθεση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Μου αρέσουν πολύ τα σημεία τα οποία αναφέρονται στο γεγονός ότι αναγνωρίζεται η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία η εθελοντική τους εργασία και, ε, γιατί χωρίς αυτή τους τη συμβολή η κοινωνία ε, θα ήταν ξεκρέμαστη. Καταλαβαίνω επίσης το γεγονός ότι αναφέρονται και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αναφέρονται οι συντάξεις. Ε, θα έχουμε και το πράσινο βιβλίο, ελπίζουμε τον επόμενο μήνα και θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Τα συστήματα τα συνταξιδοτικά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχρονισμού αν θέλουμε να είναι βιώσιμα η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας ε, θα μπορούσε να τονιστεί κάπως περισσότερο κατά την άποψή μου. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία το 80% των εργοδοτών ε, αναφέρουν ότι θα προτιμούσαν να μην προσλαμβάνουν κάποιον ηλικίας άνω των 45 ετών. Να μην σας πω, ε, δεν τίθεται καν λόγος για να προσλάβουν κάποιον άνω των 55. Ε, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθεί ε, το γεγονός αυτό ε, και να πούμε ότι θα πρέπει να έρθουν τα εμπόδια για αυτούς που εργάζονται πέραν της ηλικίας της ταξιοδότησης. Γιατί ακόμα και αυτοί που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα. Αυτό όμως το οποίο λείπει, κατά την άποψή μου, είναι η προοπτική, η διάσταση των, των δύο φύλων. Εδώ μιλάμε για μια κοινωνία ε, όπου ε, ο πληθυσμό θα γυράσει και όλο και περισσότερο, θα χρειαζόμαστε περίθαλψη, θα χρειαζόμαστε περισσότερη φροντίδα για τα παιδιά και ταυτόχρονα ε, σε αυτά τα πλαίσια οι γυναίκε αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ενό τριπλού φορτίου. Αν θα πρέπει να, να επομισθούν όλε αυτέ τι ευθύνε, θα πρέπει λοιπόν να, αναλυφθούν, να ληφθούν ισχυρά μέτρα για να υπάρξει καλύτερο καταμερισμό ε, των ευθυνών ανάμεσα στου άντρε, στι γυναίκε και στο κράτο. Ελπίζω λοιπόν να να ε, υπάρξει και κάποια, ε, να συμπεριληφθεί και η διάσταση των δύο φίλων στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά τα άλλα, σε ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω βεβαίω και θα πούν και οι άλλοι συνάδελφοι. Σα Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στα δύο λεπτά, αν είναι δυνατόν. Merci, Madame la Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Καστέξ. Χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή μου δίνεται δυνατότητα να δούμε ε, ε, αυτή την προβληματική και να κάνουμε τη συζήτηση για τη δημογραφική πρόκληση. Θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί στην προηγούμενη θητεία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Μάν, για ε, την έκθεσή του, η οποία νομίζω ότι φύγει τη συνολική προβληματική του θέματος δημογραφικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά τι διαπιστώσει του και τι παρατηρήσει του, πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε, μεγάλο μέρο και κυρίω με ενδιαφέρει αυτή η win-win ε, προσέγγιση. Δηλαδή η προσέγγιση αυτή ε, της, ε, σύμφωνα με την οποία πρέπει να υποφεληθούν όλοι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας ε, ε, χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Γιατί βεβαίω αυτό το πρόβλημα τη δημογραφική πρόκληση δεν είναι κάτι το καινούριο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα αυτό θα το βρούμε μπροστά μα. Έπρεπε να έχει ληφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Όμω τα συγκεκριμένα μέτρα ε, έχουν καθυστερήσει. Και Ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρξουν μεγάλε ανισότητε όσον αφορά ε, τι επιπτώσει ε, και οι συνέπειε θα είναι διαφορετικέ. Υπάρχει, ένα, ε, υπάρχει εδαφική διάσταση με συγκέντρωση των ηλικιωμένων ή των νέων σε ορισμένες περιοχές, στις, στις παραγωγικές και μη παραγωγικές περιοχές αν θέλετε και όλα αυτά ενδεχομένως να οδηγήσουν σε έλλειψη ισορροπίας και σε διαφορές και ως προς το κόστος αντιμετώπισης δημογραφικής πρόκλησης. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη ε, αντίληψη για τις συνέπειες. Και επίση να συνειδητοποιήσουμε ότι και η, ε, η, ε, η, ο των γεννήσεων διαφέρει ανάλογα με τι περιοχέ και ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ με τον εισηγητή στο γεγονό ότι μία πρώτη απάντηση πρέπει να δοθεί στο ερώτημα της ε, ε, οικογενειακής πολιτικής. Και εδώ πρέπει να συμβάλλουμε με, με τις συγκεκριμένες λύσεις για να ενισχύσουμε τις, ε, τον αριθμό των γεννήσεων. Αν θέλετε να τελειώνετε, λέει η πρόεδρος, γιατί έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο μιλητών. Ναι, ναι, λίγα λεπτά ακόμα. Λυπάμαι, δεν έχουμε ε, ε, λεπτά. Αν θέλετε να τελειώνετε. Ωραία, όσον αφορά το βασικό πρόβλημα, που είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Όπως ε, θα συμφωνήσετε, υπάρχει ένα πρόβλημα ανεργίας νέων, αλλά και ανεργίας ηλικιωμένων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική πολιτική ανθρωπίνων πόρων, όπου οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ε, κλείνουν τα μάτια τους απέναντι στο πρόβλημα αυτό και να ε, μην αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ε, της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων. λυπάμαι, λέει η πρόεδρος. Πέντε λεπτά ακόμα, λέει η Όχι, όχι, λυπάμαι, θα σας διακόψω. Λυπάμαι, λυπάμαι ειλικρινά, λέει η πρόεδρο, αλλά έχουμε την ψηφορία στι 9.30 και έχω έξι ακόμα μιλητέ. Ε, αυτή είναι η δυσκολία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις τροπολογίες όταν θα υποβληθούν. Ο κύριος Σέρκας έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές, αλλά δώστε της ένα λεπτό τουλάχιστον για να, για να ολοκληρώσει. Ε, μην, δεν την, δεν την ειδοποίησατε, δεν την προειδοποίησατε ένα λεπτό πριν. Ε, δώσε την ευκαιρία, ε, τουλάχιστον για λόγους ευγένεια. Να ολοκληρώσει. Μα την προειδοποίησα, την προειδοποίησα Και σα είπα σε όλου δυόμιση. Ξεπέρασε ήδη τα τρία λεπτά. Ε, νομίζω ότι είναι άδικο για του υπόλοιπου ομιλητέ. Ειλικρινά λυπάμαι ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να είμαι δίκαιη απέναντι σε όλου. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπατε. Να δώσω όμω το λόγο τώρα στην κυρία Μπάρ. Τρία πολύ σύντομα σχόλια δύσκολο να συζητάμε αυτό το θέμα. Όταν η... στην κοινωνία κυριαρχεί ένα φετίχαν θέλετε της νεολαίας και η κοινωνική διάσταση πάει πολύ πέρα από αυτό όμως. Το δεύτερο θέμα είναι η οικονομική διάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για τους κοινωνικούς πόρους, ο οποίος πρόκειται να ενταθεί στο μέλλον. Θα είναι πολύ πιο δαπανηρή η παροχή πρόνοιας και φροντίδας, θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των νέων για αυτή την κοινωνική πρόνοια. Και το τρίτο σημείο είναι η διάσταση του φύλου. Πιστεύω ότι αυτό θα φανεί και στην γνωμοδότησή μας, αλλά και τελικά στην έκθεση. Ευχαριστώ. Μιραντσότη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μωράν Σαρτιέ. Δύο βασικά θέματα. Καταρχάς, όσον αφορά την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, την διαγενειακή αν θέλετε, που αφορά την αλληλεγγύη των γενεών. Όντως, για να λειτουργήσει η κοινωνία μας πρέπει να βλέπουμε μαζί τα προβλήματα και των νέων και των ηλικιωμένων και αυτό μου άρεσε στην έκθεση, ενώ το δεύτερο που μου άρεσε είναι η σύμβαση για τα άτομα άνω των 50 ετών. Γιατί πολύ συχνά ασχολούμαστε με τους ηλικιωμένους μόνο αφού συνταξιοδοτηθούν. Όμως έχουμε και αυτό την ομάδα άνω των 50 ετών που σιγά σιγά φεύγουν από την εργασία με την ε, συνενοχή αν θέλετε των επιχειρήσεων. Τώρα, κάτι άλλο. Η επιλογή του χρόνου για τα άτομα που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, που μπορούν να επιλέγουν το χρόνο δουλειά τους. Θέλω να πω ότι για να συνεχιστεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η κατάρτιση διαβίου, Χρειαζόμαστε και κοινωνική ευθύνη επιχειρήσεων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε επίσης στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βιτσούτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα στηρίξω τις ε, ιδέες ε, του εισηγήτη η θέση του Κοινοβουλίου εδώ είναι πολύ σημαντική όσον αφορά το δημογραφικό. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, η σύμβαση για τα άτομα άνω των 50 είναι πολύ σημαντική. Και να τονίσω κάτι που, που έχουν διατυπώσει ορισμένοι συνάδελφοι όσον αφορά την κατάργηση της πρόορης συνταξιοδότησης. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν κανόνες που ισχύουν. Συνήθως κάποιοι επιλέγουν την πρόορη συνταξιοδότηση επειδή είναι μακροχρόνια άνεργοι. Οπότε το να μιλήσουμε για κατάργηση της πρόορης συνταξιοδότησης αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλη δυσαρέσκεια σε αρκετά κράτη-μέλη που έχουν τέτοιες διατάξεις. Εφόσον ε, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας αυτών των ηλικιωμένων, δεν θα έπρεπε να καταργήσουμε την προερή συνταξιοδότηση. Και όσον αφορά την οικογενειακή ζωή. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις για την αύξηση της γονικής άδειας, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχουν ακουστεί. Θέλω να βάλω την ε, εξής διάσταση στο θέμα. Ε, η αλληλεγγύη των ε, γενεών περιλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο που λέγεται δημογραφικό πρόβλημα. Ε, η γερασμένη Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους νέους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι κοινωνικές και οι οικονομικές πολιτικές και οι μακροπρόθεσμες στοχεύσεις θα πρέπει να, να θεσπίσουν κίνητρα για περισσότερες γεννήσεις ε, το λέω αυτό και ολοκληρώνω λέγοντας ότι στην περίοδο κρίσης που περνάει η Ευρώπη, κατά την οποία έχουμε περιορισμό οικονομικών πόρων, μείωση συντάξεων κλπ, θα πρέπει να μην κόβουμε, το λέω ευθέως, τα επιδόματα εκείνα τα οποία βοηθούν τα νέα ζευγάρια και τους δημιουργούν κίνητρο για α, γεννήσεις αυτό που συνέβη στην Ισπανία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα που πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, είναι κάτι που ε, νομίζω θα πρέπει να προσπαθούμε να αποφεύγεται. Όταν κόβεις ε, τα χρήματα εκείνα, τα επιδόματα για τις νέες γεννήσεις και την ανατροφή των παιδιών, δεν συμβάλλεις στο να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριος Higgins. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με την οικονομική κρίση τη σημερινή υπάρχει επίθεση στην ιδέα ότι θα έπρεπε να έχουμε συνταξιοδότηση σε λογική ηλικία και σε πολλές χώρες βλέπουμε να αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης στα 68. Μας λένε ότι πρέπει να δουλεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι επειδή μειώνεται ο πληθυσμός των νέων και επειδή δεν μπορούν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ώστε να μπορούν να παρασχεθούν ε, οι απαραίτητες φροντίδες στους ηλικιωμένους. Αυτό είναι κατάφορα λάθος. Όταν ήμουν νέος, το βασικό πρόβλημα που θα έχουμε στο μέλλον, έλεγαν οι εφημερίδες, είναι το τι θα μπορούμε να κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, γιατί θα έχουμε υπερβολικά πολύ ελεύθερο χρόνο εξαιτίας της αύξησης της τεχνολογίας. Τώρα το μόνο που βλέπουμε είναι ότι εξαιτία της βελτίωσης της τεχνολογίας είναι ότι δουλεύουμε όλοι πιο πολύ από ό,τι ποτέ και απλά αυξάνεται η ανεργία. Βλέπουμε δηλαδή ότι πρέπει να δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι να πεθάνουν. Και έχουμε έλεγχο από τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και έλεγχο και των οικονομικών πόρων από τους ε, καρχαρίες ε, και τις ε, τραπεζικές αγορές και τις καις αγορές οι οποίοι σκερδοσκοπούν λες και είμαστε καζίνο. Μήπως μπορείτε να ολοκληρώσετε εδώ, παρακαλώ. η σύγκρουση δεν είναι μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, αλλά μεταξύ της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του μεγάλου κεφαλαίου. Ο κ. Μάρκ, ευχαριστώ. Θα είμαι ε, σύντομος. Πολλά ελεύθερη. ήδη. Θα ήθελα όμως και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Μαν για αυτό το πρώτο σχέδιο, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και το οποίο αναφέρει πάρα πολλούς τομείς πολιτικής. Κάτι το οποίο θα ήθελα να πω και το οποίο πρέπει να εξακολουθήσουμε να το συζητάμε σε βάθος, είναι το σύστημα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και η διασφάλιση των συστημάτων αυτών. Βεβαίως αυτό έχει σχέση με το θέμα ε, της αντιμετώπισης ε, της μετανάστευσης και εδώ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές εξελίξεις προς τη μετα... μετανάστευση στα διάφορα κράτη-μέλη θα επηρεάσουν και το ζήτημα αυτό. Αν λοιπόν δεν βρούμε λύση στο πρόβλημα της μετανάστευσης, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε ε, αυτά τα ε, βιώσιμα και ασφαλή συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Κάτι άλλο σαν αφορά την κατάρτιση κτλ. Εδώ τα βασικά εργαλεία ε, είναι στα χέρια των κράτων μελών, αλλά η δική μας πρωτοβουλία είναι καλή και θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. έτσι ώστε να προωθεί περισσότερο το ζήτημα στα κράτη-μέλη. Ε, πριν δώσουμε το λόγο στον Τόμας Μαν, να ρωτήσουμε την Επιτροπή κατά πόσον θέλει να πει δύο λόγια. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια σύντομη παρατήρηση που Ah, yeah. Sorry. Sorry. Um, ευχαριστώ. Αυτό αφορά κάτι ε, που έχει να κάνει με το γεγονό ότι εμεί, και αφορά την έκθεση, ε, αφορά την ανακήρυξη του 2012 ε, ω το έτο για του ηλικιωμένου. Είναι εξαιρετική λοιπόν η ευκαιρία που μα δίνει η έκθεση Thomas Mann για να κάνουμε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει για την υλοποίηση αυτή τη ιδέα του Ευρωπαϊκού Έτου. Βεβαίω δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύουμε ότι ήδη από αυτό το στάδιο θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποιε ιδέε όσον αφορά του στόχου που θα μπορούσαν να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού αυτού έτους. Την Δευτέρα το Συμβούλιο θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα για την ε, ενεργό γύρενση και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιε συγκεκριμένε προτάσει, όπω ορισμένε από αυτέ που περιέχονται ε, στην έκθεση του κυρίου Τόμα Μάρτη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ που ήσασταν σύντομο. Ω κοιόδη για την ομάδα Άλντε θα αναφέρω κατηδίαν τι παρατηρήσει μου στον κύριο Τόμα Μάν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μάν για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο όπω ζητήσατε. Έθιξα απλώ ορισμένα θέματα τη έκθεσή μου προηγουμένω. Συμφωνώ με την κυρία Κόρνελίσεν. Για παράδειγμα, έχουμε πράσινη βίβλο για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και επειδή αυτά συζητούνται ξεχωριστά δεν τα έβαλα στην εκθεσή μου διότι αυτό βλέπουμε συχνά ότι παραφορτώνουμε τις εκθέσεις. Βάζουμε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα μέσα και δεν δίνουμε επαρκώς έμφαση στα πιο απαραίτητα. Συμφωνώ και με το θέμα που θίξατε για την ισότητα των φύλων. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρεται στην έκθεσή μου δύο φορές, αλλά ασφαλώς μπορεί να διευρυνθεί η αναφορά αυτή με τροπολογίες. Χαίρομαι που επίσης ε, θέσατε το θέμα αυτό της αμοιβαία εποφελούς ε, διαρρύθμισης. Επίσης συμφωνούμε για τα θέματα της παιδείας. Για την κυρία Μπάουερ τώρα είναι τεράστια η σημασία των φροντίδων για του ηλικιωμένους δηλαδή κτλ. Υπάρχουν ορισμένοι νέοι οι οποίοι τα κάνουν αυτά αφιλοκερδί, αφιλοκερδό συγγνώμη, Αλλά πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα και όπου θα ενταχθούν τα πρόσωπα αυτά μέσα και συλλέξουν εμπειρίε, βλέπετε μετά και τι πλεονεκτήματα μπορεί να έχει κανεί και από την επαφή του ως νέος άνθρωπος με τις μεγαλύτερες ηλικίε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η υποστήριξη της φροντίδας στο σπίτι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσεται το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να βγει και να πει «Α, δεν έχουμε χρήματα για να εξασφαλίσουμε τη φροντίδα». Δηλαδή, κυρία Παβά, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Ασφαλώς χρειαζόμαστε την διαβίου κατάρτιση. Πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι έχουν την εντύπωση ότι κυρίως προωθούνται οι νέοι για την κατάρτιση, την εκπαίδευση κτλ. Και όχι οι πλέον ηλικιωμένοι. Για τα προσυνταξιοδοτικά τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις δηλαδή. Εμείς στη Γερμανία προσπαθήσαμε να βάλουμε τους νεότερους όσο γίνεται πιο σύντομα στην επαγγελματική ζωή και οι ε, πιο ηλικιωμένοι να φεύγουν πιο νωρίς. Αλλά τελικά αυτό που έγινε είναι ότι χάθηκαν οι θέσεις απασχόλησης και δεν, μπόρεσαν, δεν μπήκαν δηλαδή καν οι νέοι. Αυτό πρέπει να αποφευθεί. Είναι σημαντικό και νέοι και οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ λίγες δυνατότητες επαφής. Αυτές οι ηλικιακές ομάδες χρειάζονται επίσης ελεύθερο χρόνο. Εγώ δεν θέλω να πούμε στους ηλικιωμένους ότι πρέπει να εργάζεστε, να εργάζεστε, να εργάζεστε. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι, πολύ ε, ας με επιτραπεί η έκφραση, κοτσονάτι γέροι, οι οποίοι ακόμα έχουν πολλέ δυνάμει και θέλουν και να δουλέψουν και θέλουν και να κυκλοφορήσουν. Αυτού πρέπει να του ενισχύσουμε. για την επόμενη συνάδελφο, για τον κύριο Μάτσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, ναι, είναι μία από τις απαιτήσει τις οποίες δεν ανέφερα προηγουμένως, αλλά τις τονίζω. Το έτος 2012 να οριστεί έτος των ενεργών γερατιών, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα είναι τον μεθεπόμενο χρόνο. Έχουμε την ευκαιρία, εάν μας δοθεί η πολιτική υποστήριξη, να προλάβουμε να το οργανώσουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια κοινή πρωτοβουλία. Θα ήταν ωραία δηλαδή να γίνει μια κοινή πρωτοβουλία από Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ Τόμας. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 11η Ιουνίου. Εξέταση τροπολογιών στις 13-14 Ιουλίου. 29-30 Σεπτεμβρίου η, έγκριση, η απο την Ολομέλεια. Ωραία και τώρα πάμε στην ψηφορία. Πρώτη ψηφοφορία με τις ε, κάρτες σας. Αν μπορείτε λοιπόν τις έχετε έτοιμες για να δούμε πόσοι είμαστε για να ψηφίσουμε. Πρώτον, ε, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Σχέδιο επιστολές. Ε, Ιρλανδία Water for Crystal. Ε, εργαζόμενοι στην ε, Βαλένσια και στην Καστήλη Λαμάντσα ε, που συζητήθηκαν στην ομάδα εργασία. δεν υπήρξαν ε, ε στην, ομάδα εργασία του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση ε, δεν είχαμε τροπολογίε. Μία ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται ψηφοφορία. Uh, sorry, the vote is now closed. Τώρα κλείνει η ψηφορία. And the result is 40 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. There's one member without a, a voting card. Συγγνώμη, δεν έχω την κάρτα μου. Δεν έχω την κάρτα ψηφοφορία. Να ψηφίσω λοιπόν ε, ε, ε, προφορικά. Υπέρ. Στην επόμενη ψηφοφορία. Φροντίστε να συμπεριληφθεί η ψήφο σα. Να μας το πείτε έγκαιρα. Yes, Η τροπολογία πρώτη δεν γίνεται δεκτή. Συμβασμό Α. Το επόμενο θέμα τη συμβάση. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Ε, οπότε έχουμε μία σειρά από τροπολογίε ε, μέχρι το 52 που καταπίπτουν 59 αποσύρθηκε. Συμβασμός Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε 60, 61, 62 και 58 καταπίπτουν. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64-65 ε, ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός άρχιτη ψηφοφορία κλείνει δεν πήραμε υπόψη και την δική στην ψήφο εντάξει 19, 20 υπέρ, 26 κατά, μία αποχή, δεν περνάει. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 συμβατεί με τη στην 63 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβασμός C, γάμα, υπέρ, κατά ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. The vote is closed. 26 υπέρ, 21 κατά, περνάει. 68 κατά πίπτη, 69 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβασμό D υπέρ κατά περνάει. 71, 73, 76, 77, 78 καταπίπτουν. 72 το δεύτερο τμήμα μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη στον συμβασμό D. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της 72, του δεύτερου τμήματος. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Έληξε. 20 υπέρ, 27 κατά, δεν περνάει. 74 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Έληξε. In favor. 25 υπέρ, 19 κατά, δύο αποχές, περνάει. 5 falls. 75 Γιατί εγκρίθηκε ο συμβασμός C, 80 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 81 υπέρ, κατά, περνάει 79, χωριστή ψήφος που ζήτησαν οι πράσινοι, πρώτο τμήμα, βλέπετε από το notes μέχρι το exploitation, υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Vote is closed. Although uh, 27 in favour, 20 against. Uh, that is. 27 υπέρ, 19 20 κατά περνάει. Λοιπόν, το επόμενο μέρος ε, υπέρ. Those against. Κατά. Για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Part of some... Δεύτερο τμήμα της 79. Vote is closed. Λίγοι. 23 υπέρ, 24 κατά, δεν περνάει. Συμβασμός ε, υπέρ, κατά, περνάει. Οπότε 82, 83, 84, 85, 86, 87, καταπίπτουν 88 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος. 88. Oh. That's why everybody put it Thank you. Uh, the, the vote is closed. Λίγη ψηφορία. 32 υπέρ, 14 κατά. Περνάει. Compromise F. Uh, those in favor. Συμβασμό F, σίγμα τάφ, υπέρ. Κατά. Περνάει. Οπότε όλες οι υπόλοιπε μέχρι και την 96 καταπίπτουν. Πάμε 97, υπέρ. Κατά. Περνάει. 98 υπέρ. Έλεγχος, ωραία. Άρχεται για την 97 ηλεκτρονική ψηφοφορία. The Λίγοι. 27 υπέρ, 20 κατά. Περνάει. 98 υπέρ. Κατά. Ποιες; Περνάει. 99 υπέρ. Κατά. Περνάει. Η 100 Αποσύρθηκε. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100, uh, compromise G. Those in favor. Επόμενη υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, συμβασμός G. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 34 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. 102, 104, 105, 106 και 103 καταπίπτουν. Συμβιβασμό H. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε, οι υπόλοιπε μέχρι και την 113 ε, που ε, ε, αποσύρεται, καταπίπτουν οι υπόλοιπε. Πάμε στην 115. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Συμβασμός I. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116, 117 και τα λοιπά μέχρι και την 124 καταπίπτουν. Και όσον αφορά την 125 και αυτή καταπίπτει 126. Υπέρ κατά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 126. It is closed. Κλείνει. 29 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 127 συμβατή με την 126, μάλιστα πάμε στην 127. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 Καταπίπτει, ναι, αφού εγκρίθηκε 129, 131 που είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132, 132 καταπίπτει, 133 καταπίπτει, 134 προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Πρέπει να έχετε τροπολογία μπροστά σας. 134 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135, προφορική τροπολογία, πάλι την έχετε μπροστά σα, 135 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμό J, υπέρ, κατά, Άλλη ψηφορία για αυτό το συμβασμό των Τζέι. Vote is closed. 37 uh, υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. Άρα 140, 141, 142, 143, 144, 146 καταπίπτουν. 139 μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη υπέρ 139. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος 139. Άρχεται. Vote Λίγη. 21 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Uh, Χωρίς την ψηφοφορία τώρα. Ε, μέχρι το conditions υπέρ, το πρώτο τμήμα, κατά, άρχεται η ψηφοφορία στο πρώτο σκέλος 145. is 26 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο σκέλος, υπέρ. Σα δώσω συγγνώμη, λέει πρόεδρο, είναι προφορική τροπολογία. Πρέπει να ψηφίσουμε την. Α, προφορική τροπολογία στο πρώτο σκέλος, που είναι να διαγραφεί η λέξη false μετά από, τις, ε, από την έκφραση σαφή ορισμό, clear definition of. Ζητώ λοιπόν να ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Στο προφορική τροπολογία στο πρώτο σκέλος του 145. Υπέρ, κατά, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικό έλεγχο. Προφορική τροπολογία, πρώτο σκέλο. Έληξε. 24 υπέρ, 22 κατά. Δεύτερο σκέλος υπέρ, κατά. γίνεται, δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Άρχεται ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεύτερο σκέλος. Άρχεται ψηφορία. Έκλεισε 19 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, τρίτο σκέλος. Υπέρ κατά Πάλι δεν είναι σαφής. Άρχεται ηλεκτρονικός έλεγχος, τρίτο τμήμα. το 26 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά άρχεται 149 έληξε 21 υπέρ 28 κατά Απορρίπτεται. Συμβασμός και υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε, οι επόμενες ε, τροπολογίε μέχρι και την 155 καταπίπτουν. Πάμε στην 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Πάλι ηλεκτρονικό έλεγχο, 157. Vote Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 21 κατά, 3 αποχές εγκρίνατε. Περνάμε στην 158. 160 και 161 γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη Δεκαπέντε υπέρ, τριάντα τρεις κατά. Η εκατοπέντε και εκατόν Εκατόν κομπρομάζ έλ, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά, εγκρίνατα. 163, 164, 165 και 166 καταπίπτουν. 167 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικά. Για την 167. Τέλος. 22 υπέρ, 25 κατά, 168 υπέρ, κατά, η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται, 169 υπέρ, κατά, θα το ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας. να πω ότι έχουμε ένα, μέλλον παραπάνω, ένα μέλος παραπάνω από το ΕΛΚ. Ποιος θα φύγει από το ΕΛΚ και θα ξαναψηφίσουμε για την 169. Ψηφίζετε τώρα. 25 υπέρ 22 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 170 έχουμε προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, πάλι θα το ελέγξουμε. 170 ψηφίζεται. 26 υπέρ 22 κατά 23 κατά. Μάλλον εγκρίνονται. Συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέχρι την 175 καταπίπτουν. 176 και 177 ψηφίζονται μαζί. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβασμός εν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 179 μέχρι και 182 καταπίτουν. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές,

Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά. Ξανά σηκώστε τα χέρια του. 187 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 188 υπέρ, Συγγνώμη, η 188 καταπίπτει. 189 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 καταπίπτει. Συμβιβασμός όου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέχρι την 195 καταπίπτουν, 196 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. Ψηφίζεται. «28 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται». Συμβιβασμός π υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 202-207 καταπίπτουν, 205 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 209 υπέρ, κατά, άποχες, 208 καταπίπτει. 210 υπέρ. Α, καταπίπτει. Δεν με πειράζει, είναι δική μου τροπολογία. Λοιπόν, 210 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται, 211 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 2-12 υπέρ, κατά, θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. ψηφίζεται 2-12, Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 28 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. 2.13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.17 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 2.17. Πέρας ψηφοφορίας 26 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. 2.18 υπέρ κατά. Πάλι το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 2,19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2,20 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 2.21 έχει αποσυρθεί. Συμβιβασμός Q υπέρ κατά ηλεκτρονικά για τον συμβιβασμό Q. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 13 κατά. Δεν χρειαζόταν η ψηφοφορία. 2.23 ως 2.26 καταπίπτουν. 222 ως προσθήκη στο συμβιβασμό. Υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 2.27 υπέρ, Ελέγχουμε τη 222. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 21 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. 2,28 υπέρ, κατά. Μήπως μπορείτε να ξανασηκώσετε τα χέρια σας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2,29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, θα το ελέγξουμε. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. 27 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 2.30 καταπίπτει, 2.31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβασμός R υπέρ, κατά, Άποχες. Εγκρίνεται. 2.32 2.35 καταπίπτουν. 2.36 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 2.36. Πέρας ψηφοφορίας, 26 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβασμός S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.37 καταπίπτει, 2.38 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο κοιτάξουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 6 υπέρ 40 κατά. Προφανώς δεν πρόσεχα. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στη 2.39 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.40 υπέρ, α, συγγνώμη, καταπίπτει. Καταπίπτει 2.40. Η 2.41 είναι συμβατή. 2.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.42 υπέρ, Α, θέλετε να ελέγξουμε τη 241. Ψηφίζετε παρακαλώ. 241. «24 υπέρ, 23, 24 κατά, απορρίπτεται». Αλλά καλά κάνετε που ζητήσετε ηλεκτρονική. 2.42 να είναι συμβατή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.43 ναι, είναι συμβατή. 2.43 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας το ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 24 με 24. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 2 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, το ελέγχουμε για την 6. Ψηφίζεται για την 6. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά. Πάλι δεν σηκώνετε τα χέρια σας, πώς να καταλάβω. Για την 7 υπέρ, 7 κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλά, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ίσως, μάλλον κάνω λάθος. Ψηφίζουμε για την 7. Πέρας ψηφοφορίας, 23 υπέρ, 24 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τις αιτιολογικές 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, α, 9 καταπίτη. 57 προφορική τροπολογία του εισηγητή για την διαγραφή των όρων αυτοαπασχολούμενη και ανεξάρτητη υπέρ, κατά, άποχε, πάλι δεν σηκώνετε τα χέρια σας, υπέρ για την 57 κατά, άποχες, σαφές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. 27 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Η 12 καταπίπτει, 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός τι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 18 καταπίπτουν, 19 και 20 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, ξανά υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνονται. 21 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται, 24 υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας, 21 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 καταπίπτει και η 30, 29 τώρα υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζεται. 26 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές καταπι... Ε, απορρίπτεται. 32 και 33 είναι ταυτόσιμες και μάλλον καταπίπτουν. Όχι, ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ για 32 και 33. Δεκαεννέα υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά. Πάλι δεν είναι σαφές. Ψηφίζετε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφές. 38 με 10. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 35 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 35? 35 παρακαλώ, Ψηφίσατε. 31 έναντι 17. 31 31 18, εν πάση 36 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 καταπίπτει. 40 καταπίπτει. 41 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 42 και 43 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 44 υπέρ. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. 46 καταπίπτει. 47 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, και αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, ηλεκτρονικά για την 48. Ψηφίζετε παρακαλώ. Ναι, ναι, εγκρίθηκε. Κατά λάθο είπα απορρίπτεται. Ναι, είναι προφανές. 41 υπέρ, 5 κατά. 48 εγκρίνεται λοιπόν. 49 τώρα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική. Ψηφίζετε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Εσείς τι ψηφίζετε κατά. Τέλος ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκρινή. Uh, the next one is the Beres report. Uh, Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Μπερές. And uh, the, those in favor. Για το αλφά πρώτα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, 18, 19, 20, 21 εκπίπτουν. Β, υπέρ, κατά. Θα το επαναλάβω, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25, 23, 24, αυτές εκπίπτουν. 26 υπέρ. Κατά. Ψηφοφορία ηλεκτρονική για το 26. Μία ψήφος παραπανίσια διαπιστώνουμε ότι, έχει, ότι υπάρχει του, των φιλελευθέρων του Άλντε. Μία παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Ψηφίζουμε λοιπόν ξανά. 26. Άρχεται η ψηφοφορία. 20 υπέρ, 26 κατά. Συμβαστική ε, σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έρχομαι στην 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 33 υπέρ κατά Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. ένας υπέρ 26 κατά. Ε, κατά 34 και 35 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Καλώς λοιπόν. 34 και 35. Πέρας. 27 υπέρ 20 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτή. Και αυτή η δύο ομάδα. Ναι, ε, είπα 27 υπέρ 20 κατά. Α, 35 και 36 εκπίπτουν. 37 υπέρ. Κατά. Θα χρειαστεί και εδώ επαλήθευση 37 λοιπόν. ...37, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 19 υπέρ 26 κατά. 38 έχει αποσυρθεί. 39 υπέρ. Κατά. Και εδώ θα χρειαστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 39. Αρχίζει. «20 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται». 40 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 40 τότε λοιπόν επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. 25 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα 40 και 42 εκπίπτουν, 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, θα χρειαστεί να γίνει ψηφοφορία, ηλεκτρονική ενώ, αρχίζει. 17 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45-46 Α, θέλετε λοιπόν ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε. Αρχίζει. Συμβαστική ε αρχίζει. Πέρας. 26 υπέρ 21 κατά. Εγκρίνεται. 50 τώρα. Υπέρ. Κατά. Ας γίνει λοιπόν επαλήθευση για την 50. Αρχίζει. Πέρας. 22 υπέρ 24 κατά. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά. Καλύτερα για να είμαστε ασφαλείς να κάνουμε επαλήθευση. 51 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 20 περί 26 κατά απορρίπτεται. Το αιτιολογικές σκέψεις. 1. Για να μπει η λέξη και ο θελός στο πρώτο μέρος υπέρ κατά. Ας, ας κάνουμε παλήθευση για το πρώτο μέρος της 1. Πέρας. 26 υπέρ, 20 μία ψήφι κατά. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Ναι. Δεύτερο μέρος της 1 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 2 εκπίπτει. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και προχωρούμε στην 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η 7, υπέρ, Α, η συμβαστική G, υπέρ. Δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Και εν πάση περιπτώσει παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια. Ο 45 υπέρ, μία ψυχός κατά. Αν, αν, αν σηκώνετε λοιπόν καλά τα χέρια σας νομίζω Βέβαια όλοι είμαστε κουρασμένοι, θα είναι σαφές το αποτέλεσμα και δεν θα χρειάζεται να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Η 10 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται... Συμβαστική age υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε παλήθευση Αρχίζει για την 15. Πέρας. 16 υπέρ, 31 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. 16 που έχει ζητηθεί η ψηφοφορία κατά τμήματα από τον εισηγητή. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έξι εκπίπτει. Προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία η οποία θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Αρχίζει. 41 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω την ε, κυρία Περές, εν απουσία της βέβαια, για το καλό αυτό αποτέλεσμα. Ακολουθεί Κρίστενσεν. Η 5 έχει αποσύρθει. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. σε. Συμβαστική σε γιατί δεν έχει αποσυρθεί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. πέντε. Προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Ζητείτε ψηφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20-21 εκπίπτουν, η 19 ομοίως, η 22 έχει αποσυρθεί, συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 εκπίπτει, η 26. Α, με συγχωρείτε μια στιγμή. 25 δεν εκπίπτει, 22. 25 υπέρ. 25 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 25. Πέρας. 26 υπέρ, 19 κατά και δύο αποχές. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά προτιμώ να επαληθεύσω Με ποιο τρόπο ψηφίζετε. Ο άλλο ε, συνάδελφος από πίσω σα. Είστε κατά λοιπόν, ωραία. Α, λοιπόν είναι 9 υπέρ, 37 κατά. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. θα γίνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 36. ...25 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται και μια αποχή. 37 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μόνο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική δηλαδή, για την τελική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. 44 υπέρ, 3 κατά και καμία άποχη. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και γκρίστενσεν. Έμιλι Τούρνεν για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πάμε Α, ο γραμματέας μου ζητεί λίγα δευτερόλεπτα για να βρει το σωστό έγγραφο. 29 λοιπόν, υπέρ, κατά, απορρίπτεται αλλά προτιμώ να επαληθεύσω 29. Πέρας. 23 υπέρ 23 κατά. Απορρίπτεται επομένω. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Α, εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, εγκρίνεται. Όλοι κουράζεστε, αλλά και εγώ κουράζομαι, είναι προφανές. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπή Πολιτισμού 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Α, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα τη ψήφου. 33 υπέρ, 13 κατά. Συμβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και προχωρώ στην 8 ε, της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 42 υπέρ κατά θα κάνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 42. ...26 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 λέει η πρόεδρος. Με συγχωρείτε 44. 44 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έρχομαστε 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 49. απεσύρθη 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά, Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Για την 58 αρχίζει η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 21 ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά. Πάλι δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 59 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. «21 ψήφι υπέρ, 24 κατά, απορρίτεται». Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 25 της Επιτροπής Πολιτισμού εκπίπτει, προχωρώ στην 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κάλτσορα 14 εκπίπτει γιατί καλύπτεται από την 64. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβαστική age υπέρ. Κατά. Παρακαλώ σηκώστε καλά τα χέρια. Συμβαστική age. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και <clears throat> προχωρούμε στην 77. Ε, 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Χάλτσο 10 έχει καλυφθεί 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 9 καλύπτεται 82 υπέρ κατά θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία για την 82. Πέρας. 24 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάλτσα 3 έχει καλυφθεί. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρώ στην 91. Αυτή εκπίπτει. Κάλτσα 2 υπέρ κατά Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. «28 υπέρ 19 κατά». «92 υπέρ κατά αποχές». «93 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Κάλτσορ 26. Η 18 έχει καλυφθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 καλύπτεται. Η 4 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 94. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 έχει καλυφθεί 19 πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ σηκώστε πάλι τα χέρια. 101 υπέρ, κατά. Θα κάνω ηλεκτρονική επαλήθευση. 101. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεκαεννέα υπέρ 27 κατά. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να επαληθευτεί. «19 υπέρ, 27 κατά». Απορρίπτεται. «105 υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά θα κάνω ηλεκτρονική επαλήθευση για την 108 33 υπέρ, 13 κατά. 109. Παρακαλώ σηκώστε καλά τα χέρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Υπέρ. Δεν σηκώνουν αρκετοί τα χέρια. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 πολιτισμού Έχει καλυφθεί αυτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πολιτισμού 16 έχει καλυφθεί. Η συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά απορρίπτεται 131 υπέρ προφορική κατά αποχές εγκρίνεται πολιτισμού 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πολιτισμού 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πολιτισμού 23 υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ας κάνουμε παρήθευση. Πολιτισμό 23. «25 υπέρ, 21 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Επαλήθευση λοιπόν για την M. Πέρας. 25 υπέρ 21 ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 144 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α συγγνώμη ε, εγκρίνεται πολιτισμό 21 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία 23 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική εν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148, 149 μαζί υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 150 υπέρ. Δεν εκπίπτει λοιπόν υπέρ Τις 150 κατά αποχές εγκρίνεται. Πολιτισμό 28 έχει καλυφθεί. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, Πολιτισμό 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολιτισμού α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 9. 24 υπέρ, 21 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 10. 25 ψηφί υπέρ, 21 κατά. Η 11 υπέρ, κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 13. 26 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι βεβαία. Ας κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία.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 κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές ας την επαληθεύσουμε αυτήν για την 4 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση «24 υπέρ, 23 κατά». Εγκρίνεται λοιπόν η 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία του συνόλου αρχίζει. Πέρας. 42 υπέρ, μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Τούρμεν. Κυρία Τούρμεν. Δεν έχουμε και πολλές ακόμα. Δύο, δύο. Προφορική ερώτηση πρώτα. Για τη μικροχρόνια φροντίδα. Ε, Συμβασμό σε α, υπέρ, κατά, αποχές. Ε, γκρίνεται. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6, 7, 6 υπέρ κατά όχι, όχι, ασαφής. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος στην 6. 32 um, υπέρ, 16 κατά. Συγγνώμη, ε, πρόκειται για τη δική μου έκθεση, έχω μπερδευτεί. 8 υπέρ. Δεν ψηφίσαμε στην 7, λέει η πρόεδρο. Δεν ψηφίσαμε την 7. Εντάξει, εμεί στενοχωριέσαι, όλοι κουραστήκαμε. Δεν νομίζω ότι ψηφίσαμε στην 7. Υπέρ. Υπέρ τη τροπολογία 7. 7 τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. συγγνώμη, είναι δύσκολο. Ελεκτρονικό έλεγχος στην 7. Sorry, can I just ask our administrator to get our voting list to the R group? Thank you. Εφτά. Ναι, ε, από ό,τι κατάλαβα ένα πρόβλημα με το κατάλληλο ψηφορία. Ε, δεν βοηθούν όλα αυτά. Ωραία, λίγη ψηφορία. Τι μπέρδεμα. Υπέρ 17, 26 κατά απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος στην 8. Vote closed. 20 in favor. υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Β, συμβασμός Β, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία στη 12. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά άκρη ψηφοφορία στο δεύτερο μέρος. Uh, vote Έληξε υπέρ 17 προς 29. Δεν περνάει, δεν εγκρίνεται. Ε, επόμενη, ε, βάλει χωρίς τη ψήφος υπέρ προς τμήμα. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος ηλεκτρονική άρχεται. έληξε 46 υπέρ, μία ψήφος κατά. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Και τώρα... Πάμε στην τελική. Τελευταία, τελευταία. Σχέδιο ψήφος. Έχετε όλοι το κατάργο ψηφορία, Να μην καθυστερήσουμε. My heart will stop beating. Διαφορετικά θα πάθω συγκοπή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 Favor. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 11. Άρχεται. Έληξε. 19 υπέρ, 22 κατά. Άρα απορρίπτεται. 12 ε, υπέρ, κατά. Αποχέσαι, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά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 αρχή της ψηφορίας ε, ε, για την 20, ηλεκτρονικού ελέγχου δηλαδή 20. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τέλος ψηφορίας. 17 υπέρ, 28 κατά. Πράγματι απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβασμός β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά εποχές αρχή ψηφοφορίας ηλεκτρονικής 32. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 32. Τέλος, 26 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κάποιος είπε ότι θέλει ότι δεν είναι σίγουρο για το 37. 37 λοιπόν έλεγχος. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές. Ναι, ναι, βέβαια, 44 υπέρ, 3 κατά. Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, συνολικά. Αρχή Τέλος, εντάξει υπέρ, μία αποχή και συγχαρητήρια στον σε Σας ευχαριστώ. And thanks everyone. That was a marathon. Ευχαριστώ για αυτό το μαραθώνιο ψηφοφορία. Δεν ξέρω εσεί πώ αισθανθήκατε. Εγώ πάντω είναι σαν να έχω τρέξει μαραθώνιο. We'll have um, two minute, three minute break. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την ακρόαση να ξεμουδιάσουμε λίγο. Λοιπόν, αν θέλετε να καθίσουμε. Δεν ξέρω, ε, ξεκουραστήκατε. Να πάμε τώρα στην ακρόαση. Λοιπόν, για όσους ε, θα μείνετε, αν θέλετε καθίστε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, τέλεια η συνεδρίαση, η ακροασία έχει να κάνει με τον αντίκτυπο ε, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου ε, στις υποθέσεις Viking, λαβάλ Ρούφερτ και Λουξεμβούργου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εκτός από τους βασικούς επιμελητές έχουμε και τον Τόμας Τζάνσεν, ο οποίος είναι ο εισηγητής από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Οι τρεις ομιλητές μας είναι ο κύριος Αρμάντο Σίλβα από την Επιτροπή, ο κύριος Μάξιμ Τσερούτη από την Business Europe και η κυρία Κάτλιν Πάσιερ από την ε, ε, ETUC. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Αρμάντο Σίλβα από την ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει ε, πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον προβληματισμό μας για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά αυτές τις τέσσερις υποθέσεις ε, οδήγησαν σε εκτενή συζήτηση για την ε, ε, υλοποίηση και εφαρμογή ε, της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων της 96 καθώς 7, καθώς επίσης και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα συλλογικής δράσης εκ μέρους των σωματείων. Είναι σαφές ότι απέχουμε πολύ από κοινωνική και πολιτική συνένεση όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των αποφάσεων όσον αφορά τα βασικά νομικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα ε, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αποφάσεις ε, ανέπτυξαν με, ε, με, με σαφή τρόπο τις εντάσεις που υπάρχουν όσον αφορά από τη μία τους περιορισμούς για που υπάρχουν ε, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο ε, όσον αφορά την υλοποίηση των, ε, της εσωτερικής αγοράς και από την άλλη το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και ζητούν να ξεκαθαριστούν οι κανόνες και να επιληθούν τα, εκρα, τα, εκρεμή νομικά προβλήματα. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι εθνικές κυβερνήσει άμεσα ή έμεσα, που επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα από τι αποφάσει, ήδη ανταποκρίθηκαν σε αυτή την έκκληση. Ε, ένας από τους ε, σημαντικότερους αντίκτυπους των αποφάσεων ε, ήταν οι αλλαγές νομοθεσίας στην Δανία, στη Σουηδία, στο κρατήριο της Κάτω Σαξονίας και στο Λουξεμβούργο στην Δανία και τη Σουηδία ε, εστίασαν την προσοχή του στη βελτίωση ε, τη συμβατότητα ανάμεσα στι συλλογικέ ε, διαπραγματεύσει όπω εφαρμόζονται με βάση του εθνικού κανόνε και στου ορισμού που βρίσκονται στην οδηγία για την απόσπαση. Επίση, τι συνθήκε κατά από τι οποίε τα σωματεία μπορούν να αναλάβουν δράση και να ασκήσουν αγωγή κατά μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσπασμένου εργαζόμενου. Στη Γερμανία υπήρξε η άρση βάση της υποχρέωσης ε, ε, ε, να να υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανόνες που δεν έχουν καθοριστεί ως καθολικά εφαρμοστές. Από την άλλη μεριά στο Λουξεμβούργο αναφέρθηκε, αναφέρθηκαν οι, βασικές, οι βασικοί περιορισμοί δημοσίου, δημοσίας πολιτικής, αλλά θα πρέπει να έχουν ξεκαθαριστεί όλα αυτά τα σημεία και στη χώρα προέλευσης. Όμως είναι σαφές ότι οι συνέπειες των αποφάσεων ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, των οποίων οι νομοθεσίες αποτέλεσαν ε, το αντικείμενο εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και των αποφάσεων. Όπως βλέπουμε εμείς στο ζήτημα, εδώ υπάρχουν γενικά, ε, ε, γενικά δύο ζητήματα ε, ευρύτερου ενδιαφέροντος και κυρίως όσον αφορά τις αποφάσεις Βάλκιν και Λαβάλ. Πρώτον, σε ποιο βαθμό τα σωματεία μπορούν να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς να υπονομεύεται υπονομεύονται οι οικονομικές, οικονομικές ελευθερίες όπως για παράδειγμα το δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσίας σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό το ζήτημα αφορά την ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές ελευθερίες και στα κοινωνικά θεμελιώδη δικαιώματα, ε, ε, και οι δύο πλευρές όμως ε, αποτελούν αντικείμενο διαφύλαξης από τις κοινέ αρχές του κοινοτικού δικαίου και από την οδηγία. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι έχουν το δικαίωμα να προσδιορίσουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για τους εργαζόμενους που αποτελούν αντικείμενο προσωρινής απόσπασης στην επικρατειά τους πέραν δηλαδή των ελάχιστων προϋποθέσεων και όρων που καθορίζονται στην Οδηγία 9671, χωρίς να υπονομεύεται και να υπονομεύεται ε, η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Αυτό έχει να κάνει ε, με την ερμηνεία των διατάξεων της 71 και κυρίως του άρθρου 3. Όσον αφορά την προστασία των, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των σωματείων να αναλάβουν συλλογική δράση, πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεν αμφισβητούν την αρχή ή την ουσία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το δικαστήριο αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι το δικαίωμα για ανάληψη συνολική εξωτερικής δράση είναι θεμελιώδη δικαίωμα. Επίση, επιβεβαιώνει ότι τα σωματεία θα εξακολουθήσουν να μπορούν να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν του εργαζόμενου, με την προπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο. Επίση, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων που έχει να κάνει με το δικαίωμα εργασία σε ένα άλλο κράτο μέλο. Ε, Επίση, η ελευθερία εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών είναι θεμελιώδει αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αρχές μεταφράζονται στην κοινοτική νομοθεσία έτσι ώστε να υπάρξει εγγύηση ισότιμου επίπεδου και ισότιμης αντιμετώπισης των ανθρώπων αλλά και των επιχειρήσεων. Μεγιστοποίηση λοιπόν των ευκαιριών για καινοτομία και ανάπτυξη και ταυτόχρονα προστασία των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων είτε μετακινούνται με δική τους πρωτοβουλία είτε αποστέλλονται από τον εργοδότη τους. Όμως, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων ή οι οικονομικές ελευθερίες θα πρέπει πάντα να διασφαλίζονται, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται εσκεμένα για να, υπο, για να υποβαθμιστούν οι συνθήκες εργασίας ή να ε, παραγνωριστούν ε, τα σωματεία τα οποία προασπίζονται ε, με γνήσιο τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων, ακόμα και αν πρόκειται για διασυνοριακές διαφωνίες. Αναγνωρίζοντας την σημασία των θεμάτων αυτών, ο πρόεδρος Μπαρόζο δεσμεύτηκε ενώπιον του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο 2009 ε, να προτείνει συγκεκριμένη νομοθεσία, ε, κατά προτίμηση κανονισμό, που θα υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης έτσι ώστε να επιληθούν τα προβλήματα υλοποίησης και ερμηνείας εν ώψη τη βελτίωση τη συμμόρφωση με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Όσον αφορά τη συνδιάσκεψη που διοργανώθηκε από την Ισπανική Προεδρία στο Βιέντο στις 17 και 18 Μαρτίου, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή αναγνώρισε, μετέφερε τη δέσμευση του κ. Μπαρόζου σε μια συγκεκριμένη πρόταση που είπε ότι θα υποβληθεί το 2011, αφού όμως ληφθούν υπόψη τα ευρήματα της διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβάνοντας και τους ε, ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους. Σημαντικέ εξελίξει προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η πρόσφατη δημοσίευση ε, της έκθεσης ε, με τίτλο «Μια νέα στρατηγή για την ενιαία αγορά». Η έκθεση αναφέρεται απευθεία στο πώς η αγορά και οι κοινωνικές διαστάσεις μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμοιβαία ενίσχυση ενίσχυση. Ιδιαίτερα να γνωρίζετε το γεγονό ότι για να, ε, για να είναι βιώσιμη αυτή η νέα ορμή στην εσωτερική αγορά, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα σημεία τριβή ε, που δημιουργήθηκαν στον κοινωνικό τομέα και να υπάρξει προσαρμογή των κανόνων τη ενιαία αγορά, έτσι ώστε να ληφθεί ανάγκη ε, ε του, ε, της κοινωνική, να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση αλλά και το τοπικό επίπεδο. Με βάση τι αποφάσει του δικαστηρίου, η έκθεση προτείνει να ξεκαθαριστούν οι διατάξει, να ενισχυθεί μάλλον η συμμόρφωση με τι διατάξει εξ Οδηγία 96-71 για να υπάρξει ενημέρωση για τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει των εργαζομένων, ε, καθώ επίση ε, να προβλεφθεί και το δικαίωμα κύρωση πάντα στα πλαίσια ε, τη ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων αλλά και τη ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Προτείνει η εισαγωγή διατάξεων για εγγύηση για εγγύηση του δικαιώματο ε, ε τη απεργία με βάση τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού 2679, καθώ επίση και επίσημου μηχανισμού επίλυση διαφορών, πάντα κατά εφαρμογή τη οδηγία. Ε, είναι χρήσιμο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο στοχός του κανονισμού ε, του 1998, ε, του 2679, είναι η επιβεβαίωση της αρχής ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, όμως αποκλείοντας οποιασδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο δικαίωμα απεργίας. Απαγορεύονται λοιπόν οι δράσεις που προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και επιβάλλουν σημαντικές απώλειες στα άτομα τα οποία μπλέκονται, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι δεν επηρεάζει η διάταξη αυτή το δικαίωμα απεργία. Ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση για τα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, καθώ επίση ε, ενημέρωση ε, των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Δημιουργείται λοιπόν ένα τέτοιο μηχανισμό ε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Ε, ο διαιτητή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να ζητήσει από το κράτο μέλο να άρει τα, ε, τα εμπόδια που θα έχουν εντοπιστεί και που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Εξετάζει τώρα η Επιτροπή τη αποδείξει τη έκθεση και θα ε, ε, κάνει συγκεκριμένε προτάσει για νέα ορμή στην, και νέο ξεκίνημα τη εσωτερική αγορά προ το τέλο αυτού του χρόνου. Ε, πρέπει να αναλυθούν οι επιλογέ για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων στα ευρύτερα πλαίσια ε, αυτή τη νέα όθηση προ την εσωτερική αγορά. Εξετάζονται διάφορε επιλογέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν το πεδίο εφαρμογή, τη νομική βάση, καθώ επίση και τα βέλτιστα εργαλεία, ε, λαμβάνοντα υπόψη ε, τι επιπτώσει συνθήκη Λισαβόνα και ε, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσον αφορά τον εντοπισμό του πεδίου εφαρμογή τη αναθεώρηση, εδώ ε, ε, υπάρχει, υπάρχει ακόμα μεγάλη διάσταση απόψεων. Κάτι την παρουσίαση των μελλοντικών προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη του περιορισμού που επιβάλλει η συνθήκη ε, όσον αφορά τι νομοθετικέ αρμοδιότητε, ε, κυρίω λαμβάνοντα υπόψη το άρθρο 153 παράγραφο 5 σχετικά με το δικαίωμα απεργία. Επίση, θα πρέπει να αποφύγει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσει που δεν πρόκειται να συμβάλλουν προ τη δημιουργία συνένεση ανάμεσα στου συνομοθέτε και στου κοινωνικού εταίρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 1996 συγκεκριμένη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, ε, έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη διευκρίνηση τη νομική κατάσταση και του νομικού καθεστώτο των εργαζομένων αυτών, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν. Ε, είχαν, ε, είχαν οδηγηθεί, ε, μάλλον είχαν, είχαν υπάρξει πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια. Εδώ μιλάμε για ένα πυρήνα υποχρεωτικών διατάξεων που θα πρέπει να επιβάλλει και η χώρα υποδοχής στου εργαζόμενους αυτούς. Ήταν ευφυής αυτός ο συμβασμός, γιατί από τη μια είχαμε την ανάγκη διευκόλυνσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών και από την άλλη της προστασίας των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων αυτών, αλλά και αποφυγής του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πιστεύουμε ότι αυτός ο συμβασμός ισχύει και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και στι οικονομικέ ελευθερίε συμπεριλαμβανομένη και τη κινητικότητα των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε πεπισμένοι για την ανάγκη ε, συνολική αναθεώρηση τη οδηγία. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσει για να βελτιώσουμε πτυχέ. Ε, πτυχέ όπου πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιωθούν διότι εκεί ήταν λιγότερο ικανοποιητική η εφαρμογή τη οδηγία. Ε, Όπω για παράδειγμα ε, ενημέρωση των εργαζομένων και των κοινωνικών εταίρων, δυνατότητα προσφυγής και προστασία κατά των καταχρήσεων. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να τα προσέξουμε περαιτέρω. Αυτό έχει να κάνει με τι λεγόμενε εταιρείε βιτρίνα που δεν έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα προέλευση και ε, ε, δρούν ω μέσο ε, για παράκαμψη των κανόνων που διέπουν τι εργασιακέ σχέσει στη χώρα υποδοχή. Αυτό δεν είναι καινούριο στην ομολογία ή στην ομοθεσία. Το κοινοτικό ε, δίκαιο ε, δεν μπορεί ε, να αποτελέσει, μάλλον το κοινωνικό δίκαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή τέτοιων καταχρηστικών πρακτικών, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε περιπτώσεις καταχρηστικές πρακτικές επιλογής του τόπου εργασίας με στόχο τη φοροδιαφυγή, την αποφυγή της επιβολής κοινωνικών προτύπων. Η οδηγία για τις υπηρεσίες στην τηολογική σκέψη 37 αναφέρει ότι μία απλή διεύθυνση δεν αποτελεί έδρα. Και, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη δραστηριότητα ε, για αυτή για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο κανονισμός 883 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που μόλις άρχισε να ισχύει απαιτεί ω απαραίτητη προϋπόθεση ε, ε, για να μπορέσει να εγγραφεί ε, στο, στο, στο, στο σύστημα ασφάλιση του εργαζόμενου στη χώρα προέλευση, Απαιτεί λοιπόν να ασκεί φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία αυτή. Επίση υπάρχει πρόβλημα σε περιπτώσει υπεργολαβία, όπου δεν είναι πάντα σαφέ το ποιο φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των συνθηκών που αναφέρονται ε, στι επιμέρου διατάξει. Η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τι νομικέ εξελίξει στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια ποικιλία ε, κανονισμών όσον αφορά την ευθύνη ε, και, ε, που συνοδεύονται από κυρώσει και από εργαλεία πρόληψη. Συνολικά φαίνεται ότι οι κανόνε αυτοί είναι αποτελεσματική όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους, όταν ε, η αλυσίδα υπερεργολαβίας είναι καθαρά εθνική. Αλλά ε, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ως προς την συμμόρφωση όταν ε, πρόκειται για διασυνοριακή υπεργολαβία. Αυτό δικαιολογεί λοιπόν το γεγονός ότι η Επιτροπή πρέπει να σταθεί ιδιαίτερα σε αυτές τις πτυχές που έχουν να κάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση διασυνοριακής υπεργολαβίας και θα ξεκινήσουμε μέσα το 2010 μια ευρεία μελέτη του προβλήματος αυτού οδηγία 2009 ε, του 52 για τις ε, κυρώσεις και τα μέτρα κατά των επιχειρήσεων ε, που χρησιμοποιούν εργαζομένους από τρίτες χώρες για πρώτη φορά αναφέρεται σε μηχανισμούς ευθύνης σε περίπτωση υπεργολαβίας. Δημιουργήθηκε ένας, ένας κοινός μηχανισμός για αποζημιώσεις και κυρώσεις σε περιπτώσεις τέτοιες. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το βαθμό με τον οποίο οι συνηθισμένοι μηχανισμοί επίβλεψης και εποπτείας στην χώρα υποδοχή αφορούν και του εργαζόμενου που είναι αποσπασμένοι. Η οδηγία προβλέπει ότι καλύπτονται απόλυτα από του εθνικού ελέγχου ω προ τι συνθήκε εργασία ε, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, στο βαθμό όμω που ε, αυτέ οι διατάξει περιλαμβάνονται σε αυτό τον πυρήνα των ελάχιστων προποθέσεων που, που παραθέτει η οδηγία. Όπω για παράδειγμα χρόνο εργασία, υγιεινή και ασφάλεια ε, και αμοιβή. Δηλαδή όλα αυτά που αφορούν ε, στενά, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό το τον τόπο στον οποίο παρέχεται η εργασία. Ο έλεγχο των υπολείπων συνθήκων που αφορούν περισσότερο τη συγκεκριμένη σύμβαση, όπω για παράδειγμα προστασία από την ε, απόλυση, ε, όλα αυτά θα πρέπει ε, να καλύπτονται από την νομοθεσία τη χώρα προέλευση. Πρέπει λοιπόν να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της χώρας υποδοχής που συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα των προϋποθέσεων της οδηγίας με βάση το άρθρο 3 της οδηγίας. Η δήλωση υπαριθμών 10 του Συμβουλίου δεν ε, διαφέρει από, αυτή την, ε, από, δεν διαφέρει από την αποδοχή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο δέχεται ότι η εθνική νομοθεσία, η οποία έχει περιοριστικό αποτέλεσμα στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών, μπορεί να δικαιολογείται όταν όμως υπάρχουν σαφείς απαιτήσει που έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, αλλά ε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αναλογικά απαραίτητα και ε, να μην διασφαλίζεται και καλύπτονται από του κανόνε που ισχύουν στη χώρα προέλευση. Τέλο, ε, ε, η επιλογή της, νομοθε... Ε, η επιλογή της νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει να κάνει με το, πρόβλημα, με το προσεπίληση πρόβλημα. Ε, οι κανονισμοί λοιπόν καταρχήν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, ε, γενικά ε, καλύτερα έναντι των οδηγιών γιατί παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τη νομική ασφάλεια για όλους τους ενδιαφερομένους. Όμως η συνθήκη επιτρέπει τη, και την χρησιμοποίηση σε άλλα στις οδηγίες όταν στηρίζεται στο άρθρο 352 πρώην εκεί όπου αναφέρεται η ομοφωνία στο Συμβούλιο και η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Ανάλογα λοιπόν με την θεώρηση, μπορεί να εξεταστεί ε, και η περίπτωση οδηγίας. Ε, υλοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε προπροσκευαστική εργασία για μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, ανεξάρτητα με τη νομική βάση ε, που θα αποτελέσει αντικείμενο επιλογής, θα συμπεριλάβει διάφορες μελέτες αξιολόγησης, ε, σχέδια κτλ. Επίσης, εξ αξιολόγηση του αντικτύπου για τις κοινωνικές και νομικές πτυχές ξεκίνησε το 2009 όσον αφορά την οδηγία. Και τα πρώτα αποτελέσματα περιμένονται στο πρώτο ε, τρίμηνο αυτού του έτου. Ε, η αξιολόγηση αυτή γίνεται με την υποστήριξη του πολιτικού σχεδίου που πρότεινε το 2008 το Κοινοβούλιο. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει τι δυσκολίε ω προ την ερμηνεία τη οδηγία. Όπως για παράδειγμα η εφαρμογή της έννοιας ε, των, ε, των διατάξεων δημόσιας πολιτικής, ε, η, η κάλυψη ελάχιστων αποδοχών και το πώς μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Η Επιτροπή θα εξακολουθεί στην εργασία της για να μπορέσει να, υπά... για να, μπορέσει να επιτευχθεί συνένεση και στα πλαίσια αυτή τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασία με την εξή αποστολή. Αξιολόγηση τη σκοπιμότητα ενό συστήματο ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών που θα διευκολύνει τι επαφέ ανάμεσα στι εθνικέ διοικήσει. Μελέτη σκοπιμότητα για τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συνεργασία ανάμεσα ε, στι επιθεωρήσει εργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη αδήλωτη εργασία. Ξεκίνησε λοιπόν μια τέτοια πρωτοβουλία το 2009 και και τα αποτελέσματα αυτή τη πρωτοβουλία τα περιμένουμε ε, στο τελευταίο τρίμηνο του έτου αυτού, του 2010. Επίση, υποστηρίξαμε πέντε διεθνικά σχέδια ε, ε, και καθώ και διάφορε προσκλήσει υποβολή προτάσεων 2009, έτσι ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στενά σε θέματα απόσπαση εργαζομένων να μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίε και βέλτιστε πρακτικέ. Παρόμοιε προσκλήσει υποβολή προτάσεων θα συνεχίσουν το 2010, πάλι με τη βάση των πιλωτικών σχεδίων που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι, ελπίζω να ξεκαθάρισα το γεγονό ότι η ανάγκη για την εισαγωγή διασαφηνήσεων και για να, ε, δώσουμε απαντήσει ε, στα θεμητά ε, ερωτήματα των εμπλεκομένων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζω ε, στα πλαίσια της προόδου του εσωτερικού προβληματισμού και εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να απάντησα σε τις ερωτήσεις και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα να διασαφηνίσω και άλλα σημεία στα οποία τυχόν δεν απάντησα. Ευχαριστώ. Θα περάσω στην Κατλέν Πασχή που είναι η υπεύθυνη γραμματέα για την απόσπαση εργαζομένων της ΕΤΟΚ, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα βασικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και άλλα στοιχεία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Έχετε μπροστά σας αντίγραφο των ε, διαφανειών, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να δείξουμε τώρα τις διαφάνειες και ίσως δεν κρατήσει ακριβή σειρά των διαφανειών για να μπορέσω να τηρήσω τους χρονικούς ε, περιορισμούς. Να πω ότι μαζί με το σώμα σας είχαμε ανησυχίες ε, για το πώς τέθηκε σε ισχύ, για το πώς εφαρμόζεται, αλλά και γενικά για την ίδια την νομοθετική πράξη. Να πω ότι για εμάς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εσωτερική αγορά για την οποία μιλάμε, όταν μιλάμε για συλλογικές διαπραγματεύσεις, για αποσπάσεις κτλ, δεν είναι αυτός σκοπός είναι ένα εργαλείο για να επιτύχουμε πρόοδο για όλους τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Και υπό αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα έγγραφα. Ας δούμε τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου. Στις διαφάνειες χρησιμοποίησα όρους ποδοσφαιρικούς. Ειδικά στην περίπτωση Viking έχουμε σκορ 4-1 υπηρεσίες κατά εργαζομένων. Γιατί, γιατί και είναι ενδιαφέρον αυτό έχοντας ακούσει και τον κύριο Σίλβα ότι θέτει το ερώτημα ακριβώς όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς. Υπάρχει ιεραρχία. Το ερώτημα για τον κύριο Σίλβα είναι τα συνδικάτα και τα κράτη-μέλη όταν κάνουν κάτι δεν πρέπει να υποσκάτουν την αγορά. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αν ήταν ισορροπημένη η αντιμετώπιση του δικαστηρίου θα έπρεπε να, έπρεπε να υπάρχει και το ερώτημα όταν έχουμε μεταφορά εργαζομένων ή εταιριών δεν θα έπρεπε να φροντίζουν να μην υποσκάπτουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή θα ήταν μια ισορροπία η οποία λείπει αυτή τη στιγμή από τις δικαστικές αποφάσεις. Μας ρωτάτε για τις συνέπειες των συλλογικών δραπαγματρεύσεων. Βλέπετε στις διαφάνειες τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε εμείς ως συνδικάτα όταν αναλαμβάνουμε συλλογική δράση για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους σε περιπτώσεις όπου έχουμε διασυνοριακή διάσταση. Και αυτό εύκολα μπορεί να γίνει σήμερα στην Ευρώπη. Κάθε φορά όμως που κάνουμε κάτι τέτοιο υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε στο δικαστήριο και όποια εταιρεία μπορεί να βρει ένα επιχείρημα ότι υπάρχει διασυνοριακή διάσταση προβάλλει το επιχείρημα αυτό και το επιχείρημα του κινδύνου για την ελευθερία μετακίνησης της εταιρείας. Αυτό ήταν το επιχείρημα για την ε, για το Βρετανικό Συνδικάτο που προσπάθησε να αντιταχθεί στην British Airways και σε άλλες υποθέσεις που κατέληξαν στο δικαστήριο. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και εμπρό. Θεωρούμε ότι η εσωτερική αγορά είναι σημαντική και τη στηρίζουμε. Πρέπει όμως να οικοδομήσουμε και την εμπιστοσύνη. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όμως πρέπει να υπάρχει σαφής δήλωση του τι ισχύει για τους εργαζομένους στην αγορά. Υπάρχουν οδηγίες και αναγνωρίζουν την ανάγκη προστασίας. Και εδώ πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ προστασίας και προστατευτισμού. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Άλλο ερώτημα είναι εμπόδιο οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η συλλογική δράση. Σε τι βαθμό είναι εμπόδιο. Νομίζω ότι δεν βλέπουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Άρα εμείς έχουμε πολύ σαφείς απόψεις για το τι πρέπει να γίνει, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Θεωρούμε ότι η ισορροπία αυτή τη στιγμή είναι λανθασμένη και θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση σε επίπεδο συνθεκών. Εμείς μιλάμε για ένα πρωτόκολλο κοινωνικής πρόοδου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θα έπρεπε να είναι κατά. Εξάλλου η κοινωνική πρόοδος αναφέρεται και στη συνθήκη. Άρα πρέπει να υπάρξει ερμηνεία των συνθήκων και να αναφερθεί ότι οι συνθήκες έχουν αυτό το στόχο. Άρα η εσωτερική αγορά δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με το αν αυτό που κάνουν τα συνδικάτα υποσκάπτει την εσωτερική αγορά, αλλά και το κατά πόσο οι επιχειρήσεις υποσκάπτουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο εργαζόμενος δεν είναι υπηρεσία. Μια υπηρεσία παρέχει, μια εταιρεία μάλλον παρέχει υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μπορεί να τις παρέχει οπουδήποτε, όμως πρέπει να υπάρχει και νομικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους. Η οδηγία για τις υπηρεσίες, η οδηγία για τις αποσπάσεις, και βεβαίως από εκεί και πέρα έχουμε και την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος Μόντι πρόσφατα έγραψε μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση την οποία μελετούμε ενδελεχώς. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζει το πρόβλημα της νομιμοποίησης της αγοράς όμως διαπιστώνουμε ορισμένα προβλήματα στα επιχειρήματά του όταν μιλάει για τις οικονομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνει καλά ποια είναι τα προβλήματά μας με την οδηγία για τις αποσπάσεις. Και δεν εξέτασε σε ποιο βαθμό θα μπορούσε η αναθεώρηση του κειμένου να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης θα θέλαμε να προτείνουμε ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες που είναι παρόμοια με αυτή για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών. Όμως και η οδηγία για τις αποσπάσεις δεν είναι διαφορετική από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εκεί να έχουμε ένα σύστημα επίλυσης διαφορών και να μην υπάρχει αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που αμέσως μας επιτίθεται κάθε φορά που λέμε ότι θα αναλάβουμε δράση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για εμάς αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουμε επίσης την δυνατότητα στο παράγωγο δίκαιο να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων βλέπετε και άλλες προτάσεις που έχουμε για την οδηγία αυτή καθ' αυτή. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, πάντως μόλις ολοκληρώθηκε η έκθεση εμπειρογνωμόνων της ΕΤΟΥΚ που αναφέρει διάφορα πράγματα σχετικά με το νομικό πλαίσιο κτλ. Θα σας τα στείλω στα αγγλικά και στα γαλλικά. Χτες ολοκληρώθηκε αυτή η έκθεση. Τώρα, ο κανονισμός που ανακοίνωσε η Επιτροπή μπορεί να λύσει τα προβλήματά μας. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Όμως επικεντρώνεται στην υλοποίηση και την εφαρμογή. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, η κοινωνική εταίροι μας, η FIAC και η WW, και αυτοί προσπαθούν στο πεδίο των κατασκευών να βελτιώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όμως, ακούγοντας τον κύριο Σίλβα, αλλά και τις άλλες συζητήσεις που είχαμε με την Επιτροπή, θεωρούμε ότι δεν επιλύονται έτσι τα προβλήματά μας με την οδηγία, η οποία είναι οδηγία μέγιστων ορίων. Μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ερμηνεύσουμε στο πλαίσιο της συνθήκης. Μπορούμε να προσφέρουμε προστασία πέρα από αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις της οδηγίας για τις αποσπάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν επιλύεται με τον κανονισμό. Επίσης, ο κανονισμός καλύπτει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Για παράδειγμα, είμαστε υπέρ ενός συστήματος κοινή ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τα εθνικά συστήματα δεν μπορούν να καλύψουν τις διασυνοριακές υποθέσεις. Όμως, όταν περνάμε σε πιο ευαίσθητα θέματα, θεωρούμε ότι θα είναι εξίσου δύσκολη η έγκριση αυτού του κανονισμού όσο και με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποσπάσεις. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι θα χρησιμεύσει τόσο πολύ ο κανονισμός. Εν πάση περιπτώσει θα εξετάσουμε προσεκτικά την πρόταση της Κομισιόν και ελπίζουμε ότι κάποιες από τις ανησυχίες της ΕΤΟΚ αλλά και του Κοινοβουλίου πρόσφατα θα ληφθούν υπόψη. Τέλος, κάποια πράγματα σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι η, έκθεση, η υπόθεση Ρούφπερ είχε καταστρεπτικές συνέπειες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι ότι καταρχάς η απόφαση είναι κατά του πνεύματος της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες και σίγουρα είναι και αντίθετη με το γράμμα της σύμβασης του ILO του 1994 που την έχουν επικυρώσει 10 κράτη-μέλη. Και δεν μας λέει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή πώς θα μπορέσουν να συνδυάσουν την απόφαση του δικαστηρίου αυτά τα κράτη-μέλη με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη σύμβαση του ILO. Όμως η σύμβαση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί προστατεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα, υποθέτω ότι ορισμένα θα τα ξανακούσουμε Γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε και για την ε, συνεργασία μας με τους εργοδότες επί του θέματος. Νομίζω ότι είχαμε επικοδομητική συζήτηση τον τελευταίο χρόνο και με ευχάριστη ατμόσφαιρα αποφασίσαμε ότι συμφωνούμε να διαφωνούμε, τουλάχιστον για τα πιο σημαντικά θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διακόψουμε τις συζητήσεις, ειδικά σε ευρεία θέματα όπως η, η κινητικότητα. Και σίγουρα είναι σημαντική η συνεργασία και συζήτηση των κοινωνικών εταίρων, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία επί των βασικών θεμάτων που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. από την Business Europe, την ε, Συνομοσπονδία των ε, Εργοδοτών στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο κύριε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Τσερούτη, που μας προσκαλέσατε για να σχολιάσουμε τις τέσσερις αποφάσεις του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η έκθεση αναφέρεται στις αποφάσεις αυτές και στις αμφιλεγόμενες. Δείχνει και που συμφωνούμε αλλά και που έχουμε διαφορές απόψεων. Στις 19 Μαρτίου ολοκληρώσαμε την έκθεσή μας αυτή και από τότε ακούσαμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθεί για την απόσπαση εργαζομένων δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο και το ίδιο έχει υποστηρίξει και ο κύριος Μόντι στην έκθεσή του. Πιστεύουμε ότι η έκθεση είναι μια ισορροπημένη συμβολή στην ε, συζήτηση για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας περί αποσπάσεως εργαζομένων. Έχω φέρει και μερικά έντυπα, αντίτυπα δηλαδή, της ε, έκθεσης αυτής. Ήταν μακρά η διαδικασία, όπως είπε και η Κατλίν προηγουμένως, αλλά πραγματικά μελετήσαμε ε, ενδερεχώς όλα τα θέματα. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θα ήθελα τώρα να φωτίσω ιδιαίτερα και όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρώτα, η αρχή ελεύθερη διακίνηση προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί σωστά. Πρέπει να καταπολεμηθεί ο προστατευτισμός. Δεύτερο, η κινητικότητα των εργαζομένων και των εταιριών στην ενιαία αγορά. Είναι βασικό στοιχείο για την περαιτέρω οικοδόμηση της Ευρώπης και από οικονομικό και πολιτικό και ε, για οικονομική πολιτική και κοινωνική σκοπιά. Επίσης για να διατηρηθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση να υπόκειται στους ίδιους κανόνες και να μην υπάρχει διάκριση. Και τέλος η οδηγία αποσπάσεως εργαζομένων που αναφέρεται εν τέλει σε 0,4% του εργαζόμενου δυναμικού στην Ευρώπη πρέπει να εφαρμοστεί με καλύτερο τρόπο. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία συμφωνούν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι. Τώρα εδώ σήμερα προσερχόμαστε για να εκφράσουμε τις απόψει μας για το τι θα πρέπει να γίνει ω επόμενο βήμα. Πρώτα όμω, θα, ήθελα να επανέλθω στο τι έχετε κάνει εσεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η Ευρωβουλή. Στην τελευταία έκθεση που ε, εγκρίνατε τον Οκτώβριο του 2008 είναι για τι ε, συλλογικέ συμβάσει και είπατε τότε ότι μια μερική αναθεώρηση της ε, οδηγίας περί αποσπάσεων εργαζομένων δεν θα πρέπει να αποκλείεται εάν θεωρηθεί απαραίτητο μετά από ανάλυση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Συμμετέχοντα στην ακρόαση αυτή, εμείς θέλουμε να καταδείξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει λόγο να αναθεωρηθεί η εν λόγω οδηγία. Πρώτος λόγος, το δικαίωμα απεργία και συλλογικών συμβάσεων διατηρείται. Κάτι που όπως στις περιπτώσεις Λαβάλ και Βάικινγκ ε, έχει αγνοηθεί. Αναγνωρίζεται όμως για πρώτη φορά το δικαίωμα της απεργίας ως θεμελιώδες δικαίωμα. Από τότε όμως υπήρξαν και άλλες ε, εξελίξεις από τον Δεκέμβριο του 2009 που ε, μπήκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και δίνει περιλαμβάνει τον χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων ως πρωτογενές δίκαιο και είναι σημαντικό να εκτιμηθεί και να αναλυθεί ποια είναι η νομική συνέπεια αυτής της εξέλιξης, διότι εν τέλει γύρω από τα θέματα αυτά και γύρω από τους προβληματισμούς αυτούς που θέτει και η Ευρωπαϊκή ΓΕΣΕΗ, η ΙΤΑΚ, αυτά είναι πρέπει να συζητηθούν σήμερα. Και νομίζω ότι θα επιληθούν με τον τρόπο αυτό πολλά, πολλές από τις ανησυχίες. Σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού, το δικαίωμα απεργίας δεν είναι απόλυτο. Απόλυτα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, η απαγόρευση βασανιστήριων κτλ. Αυτά δεν μπορούν να περιορίζονται. Όμως το δικαίωμα στην απεργία πρέπει να ασκείται αναλογικά. Γιατί χωρίς τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να περιορίσει άλλες ελευθερίες σημαντικά. Και αυτό ισχύει και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα το δικαίωμα της ε, Ελευθερία έκφραση το οποίο σα απασχολεί ιδιαίτερα εσά εδώ τους Ευρωβουλευτέ. και αυτό πρέπει πάλι να ασκείται με τρόπο αναλογικό. Οι ε, αποφάσει του δικαστηρίου δεν εφευρίσκουν τον τροχό, δεν πρωτοπορούν. Η αναλογικότητα στην άσκηση της ε, συλλογικής δράσης είναι απαραίτητη. Και υπάρχουν και στις νομοθεσίες των χωρών μελών ορισμένες νομοθετικές ε, Ορισμένε νομοθεσίε, μάλλον που όπως είπα και μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων με την ΙΤΑΚ δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε μια κοινή η άποψη. Θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και θεμελιωτών δικαιωμάτων. Αλλά τελικά δεν καταλήξαμε σε κοινέ διατυπώσει. Και ο λόγο είναι ότι για μα ήδη σήμερα οι οικονομικέ ελευθερίε είναι περιορισμένε σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, υπάρχουν εθνικοί κανόνες και η διασύνδεση μεταξύ αυτών των κανόνων οδηγεί εν τέλει στο ότι η άσκηση των ελευθεριών αυτών πρέπει, περιορίζεται σημαντικά. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό που είπε είναι ότι το δικαίωμα συλλογική δράση πρέπει να ασκείται και αυτό ε, αναλογικά. Άρα υπάρχουν αμοιβέ παραχωρήσει. Αυτό δεν αποτελεί τίποτα το εξαιρετικό. Για να φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό διότι όπως είπα και οι δύο πλευρές πρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους με τρόπο αναλογικό. Τα μέτρα που λήφθηκαν στις θυγόμενες χώρες μέλη για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου δεν θίγουν νομίζω τα δικαιώματα των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν αμφισβητούνται τα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων των ε, χωρών αυτών. Για παράδειγμα, η ε, απόφαση Λαβάλ λαμβάνει υπόψη της, ε, τη Σουηδική νομοθεσία, όπου δεν υπάρχουν οι προβλέψεις που υπάρχουν αλλού για συλλογικέ συμβάσει κ.ο.κ. Είπε ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυτά και στις αποσπάσεις εργαζομένων. Υπήρχε λοιπόν έλλειψη διαφάνειας, η οποία τώρα, ε, η κατάσταση αυτή μάλλον τώρα βελτιώνεται. Τα μέτρα που λαμβάνονται ωστόσο ε, δεν φύγουν το σύστημα συλλογικών συμβάσεων στην Σουηδία. Επιτρέπεται, επιτρέπει την ερμηνεία των αποφάσεων. Η οδηγία αποσπάσεων των εργαζομένων θεωρούμε εμεί ότι δεν είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί. Αυτό είναι το πιο βασικό που θέλω να πω σήμερα. Γιατί εξασφαλίζει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην υπερεθνική ε, προσφορά υπηρεσιών και ταυτόχρονα επαρκή ε, προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Καθορίζει έναν πυρήνα κανόνων που οφείλουν να σέβονται οι επιχειρήσεις εάν αμφισβητούσε τους ε, υφιστάμενους κανόνες τότε θα υπήρχε θα, ε, ήταν εμπόδιο για την μετακίνηση των επιχειρήσεων και εργαζομένων. Κανόνες οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζονται το ίδιο. Δεν υπάρχουν διαφορές δηλαδή για τις επιχειρήσεις. Και αυτός είναι και ο στόχος της οδηγίας, δηλαδή να περιοριστεί η χρήση αυτών των ε, ε, κανόνων ίσης μεταχείρισης στις ε, επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες προχωρούν σε απόσπαση εργαζομένων και προσφέρει επαρκή προστασία στους αποσπασμένους εργαζόμενους καθορίζοντας ξεκάθαρα τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται και βεβαίως και, τους ελάχιστες, και τις ελάχιστες αμοιβέ που είναι ασύνηθες όπως γνωρίζετε στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λόγο στις αμοιβέ των εργαζόμενων. Αυτά είναι υπόθεση των χωρών μελών και των συλλογικών συμβάσεων. Αλλά επειδή είναι οδηγία συντονισμού και όχι εναρμόνισης, το θέμα της ε, αμοιβή έχει αναφερθεί. Θεωρούμε ότι δεν επηρεάζεται η ισορροπία αυτή από τι αποφάσει του δικαστηρίου και αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση. Ο πυρήνα των κανόνων μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη στα διάφορα εθνικά πλαίσια η δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητο για να υπάρξει διοικητική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και καλύτερη ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζόμενων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αυτό είναι μια προϋπόθεση για να υπάρξει καλύτερη βελτιωμένη εφαρμογή της οδηγίας και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος για να βελτιωθεί οποιαδήποτε μέτρα εφαρμογή της οδηγίας, αυτό είναι σημαντικό για μας, δεν θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει σε υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και γνωρίζουμε ότι υπάρχει και σαφή νομολογία του δικαστηρίου σχετικά με ποια μέτρα μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά και ποια όχι. Εν συμπεράσματι, είναι αληθές ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τόνισαν ορισμένα προβλήματα που διαπιστώνονται στις αποσπάσεις εργαζομένων, αλλά οι θυγόμενες χώρες μέλη έλαβαν, ανέλαβαν δράση για να βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας, χωρίς να αμφισβητήσουν τα συστήματα συλλογικών συμβάσεων των ίδιων των χώρων μελών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Ευρωβουλή θα συμφωνήσει με, με εμά ότι δεν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της ε, οδηγίας απόσπαση εργαζομένων και ότι θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος για να βελτιώσουμε τη διοικητική συνεργασία, να βελτιώσουμε την ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζομένων, που όπως είπα αποτελεί την προϋπόθεση για την συμμόρφωση. Δεν αναφέρθηκα σε ορισμένα από τα θέματα που θέσατε στι ερωτήσεις σας, αλλά είμαι βεβαίω στη διάθεσή σα για να σα απαντήσω εάν επιθυμείτε να τι θέσετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και συμπληρωματικές ερωτήσεις και ερωτήσεις follow-up. Πριν να σας δώσω το λόγο, σας παρακαλώ να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί θα ήταν χρήσιμο για τη συζήτηση. Έχουμε τους τρεις ομιλητές που θα μπορούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον πρώτο ομιλητή. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Λούντβιξον. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν την ε, τόσο ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, Βίκιν, Λαβάλ και Ράφερτ ε, συζητήθηκαν εκτενώς ε, μετά την έκδοσή τους. Και πρέπει να σας πω ότι πάντα μου προξενεί έκπληξη η επιχειρηματολογία συγκεκριμένη. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στην εξή κατάσταση. αντιμετώπισαν λοιπόν αυτές τις απειλές στα σωματεία ε, και, κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, εδώ μιλάμε για παραβίαση ε, ε διατάξεων ε, του ε, Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έχουμε δηλαδή εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους εργοδότες και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν αποδοχές που, δεν που απέχουν πάρα πολύ από οποιαδήποτε έννοια δίκαιης αμοιβή. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι για πολλά χρόνια στη Σουηδία ασχοληθήκαμε με τα ζητήματα αυτά και εγώ έχω ε, εμπειρία. έβλεπα όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους εκμεταλλεύονταν ε, όλοι αυτοί οι εργοδότες. Ε, πρόκειται λοιπόν για, για κοινωνικό ντάμπινγκ και για τίποτα άλλο. Εδώ τώρα μιλάμε για την Οδηγεί αυτή, η οποία υποτίθεται προστατεύει του εργαζόμενου και όμω τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Όταν, όταν υπάρχει ε, περιορισμός όσον αφορά την ε, δράση και επιρροή των σωματείων. Αυτή τη στιγμή στη Σουηδία δεν μπορούμε καν να απαιτήσουμε την ασφάλιση των εργαζομένων, ε, την ε, εφαρμογή της αρχής ε, ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Προφανώς λοιπόν πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις. Θέματα στα οποία δεν, αναφέρ, δεν, θέματα στα οποία δεν κάλυψε και η νομολογία. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω όμως, και απευθύνομαι στην Business Europe και στην Επιτροπή. Πραγματικά θέλετε να ασχοληθείτε με το πρόβλημα αυτό. Γιατί εδώ έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσα ε, σε σοβαρέ και λιγότερο σοβαρέ εταιρείε. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει ο θεμητό ανταγωνισμό, αλλά υπό ισότιμε συνθήκε και προποθέσει. Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση του, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, Παγκόσμιου και να την εφαρμόσουν. Και τώρα η νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση. Μα είναι σωστή αυτή η Μήπως λοιπόν πρέπει να, να, πάμε με τις χώρες που δεν θέλουν τη σύμβαση, π.χ. Αλβανία, Νότια Κορέα και Ζιμπάμπουε και πολλές ακόμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και αν θέλουμε να ακούσουμε και απαντήσεις στις ερωτήσεις, σας παρακαλώ, μπορείτε να είστε πάρα πολύ σύντομοι και να κάνετε συγκεκριμένε ερωτήσεις. 1,5 λεπτό θα ήταν τέλειο. 1,5 λεπτό το πολύ σας παρακαλώ δεν θα σας χρονομετρήσω, αλλά σας παρακαλώ, μπορείτε να, κρατήσετε να μείνετε σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Κύριος Κρίτας, Κρίστης, αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όταν η Δανία άλλαξε τους κανόνες της, λόγω του γεγονότος ότι ε, υπήρξε αυτή η απόφαση ε, του δικαστηρίου έναντι του μοντέλου εργασίας. Ε, και θέλω να ρωτήσω, της Δανίας, και θέλω να ρωτήσω τις εξής ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ε, σας κατάλαβα καλά, οι κανόνες της ιστορικής αγοράς με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν ε, είναι πλέον ε, δεν ε, ε, υπεράνω του δικαιώματος για συλλογική δράση των εργαζομένων. Δηλαδή θέλω να πω, εάν ένας αποσπασμένος εργαζόμενος ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου ε, εργάζεται κάτω από χειρότερε συνθήκε από ό,τι, από εργάζονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη χώρα. Τι γίνεται τότε. Σας ρωτώ. Γιατί, ε, όπως σας είπα, υπέστη επίθεση το, ε, το μοντέλο ε, της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μιλητή. Σας ευχαριστώ. Εν είδη προημίου, θέλω να σας πω ότι είμαι αρκετά ε, ε, ηλικιωμένο και έχω δει ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, πολύ, ευχαρι... πολύ ευτυχισμένα ακόμα και πριν από τη συνθήκη τη Ρώμη. Είμαι δάσκαλος και έχω συνεργαστεί με συναδέλφους μου από όλη την Ευρώπη. Δεν είχαν προβλήματα. Ε, και πριν την εσωτερική αγορά. Άρα δεν καταλαβαίνω εδώ περί τίνο πρόκειται. Τώρα, εδώ μιλάμε για, για, για, για συλλογική δράση και όχι για άτομα επιμέρους. Ε, βρεθήκαμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται ε, σε, ε, παίρνοντας μισθό μικρότερο από τον κατώτερο μισθό των συγκεκριμένων χωρών. Από ό,τι κατάλαβα όμως, ο κατώτερος μισθός είναι νόμος στις, στις χώρες αυτές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το δικαστήριο παίρνει μια απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με, τον, με την νομοθεσία των χωρών αυτών. Τι θέλουμε δηλαδή να προωθήσουμε τις μαζικές μετακινήσεις των εργαζομένων σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε σε τελευταία ανάλυση, ανάλυση να οδηγηθούμε στην ε, διάλυση και στην καταστροφή ε, των ε, κρατών μελών, των, των επιμέρους κρατών μελών. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κυρία Βιγκερέιδο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Και ε, έχω ορισμένα ερωτήματα, τα οποία είναι ερωτήματα επί της ουσίας, που δεν απαντήθηκαν. Ούτε από τη συνθήκη, ούτε από την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Και ούτε φυσικά και στις απαντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί κοιτάξτε, ποιο είναι το διακύβευμα εδώ. Από τη μια έχουμε τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και από την άλλη τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και ε, υπάρχουν διαφορετικές εφαρμογές της νομοθεσίας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι τελευταία ανάλυση η αρχή των ε, ίσων αποδοχών τη προάσπιση, αν θέλετε, ενό ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση. Και όχι ε, μόνο μέσω του κοινωνικού ντάμπινγκ, το οποίο σίγουρα ε, γίνεται με το πρόσχημα αυτή την απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά όχι μόνο λοιπόν μέσω του κοινωνικού ντάμπινγκ, όπως σας είπα, αλλά και μέσα από την έλλειψη ε, κοινωνικής ασφάλισης των ανθρώπων αυτών. είτε χρησιμοποιώντα ε, την ε, συγκεκριμένη οδηγία για την απόσπαση, είτε ερμηνεύοντα τι διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα. Και μάλιστα θα έλεγα, αν εξετάσουμε σε βάθος αυτή την προβληματική, ε, θα, ο μοναδικό τρόπος επίλυσης του προβλήματος θα ήταν αναθεώρηση της συνθήκη Λισαβόνα. Λέγοντα ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν μπορούν να τίθεται υπό αμφισβήτηση μέσω ε, τη αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ή τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ο ελεύθερο ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των επιχειρήσεων έχουν κάποια όρια. Και δεν μπορούν που λόγο να θέτουν σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα, τα επιμέρου δικαιώματα των πολιτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μα αυτά είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται συνθήκη και δεν αναφέρονται. Και εφόσον δεν αναφέρονται, δυστυχώ έχουμε αυτή την κατάσταση όπου υπάρχουν ποικίλε ερμηνείε ερμηνείες που πάντα είναι ει βάρο των εργαζομένων. Τώρα βεβαίω και δεν μπορώ να δεχθώ τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε εδώ. Δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η οδηγία ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Δεν δέχομαι κάτι τέτοιο και βεβαίως δεν δέχομαι αυτό το οποίο ακούσαμε. Ή μάλλον δεν δέχομαι ότι γενικά δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ ε, πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στου κοινωνικού εταίρου, και από ό,τι άκουσα και από την Business Europe τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, ε, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην ανάληψη μέτρων και να, ε, και να υποβάλει πρόταση έτσι ώστε να, το, να τεθεί ε, τέλος ε, στο κοινωνικό ντάμπινγκ για να προασπίσει τα δικαιώματα των ασθενέστερων, δηλαδή των εργαζομένων. Διαφορετικά ας πάψουμε να μιλάμε για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ας πάψουμε να λέμε ότι ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι χώρες της Ασίας, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. κύριος Φάμπρεχ το λόγο. Συμφωνώ με τα επιχειρήματα της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Να σας πω ότι το 1979 δημιουργήθηκε ο ILO, το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασίας και το δικαίωμα στην απεργία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις δημιουργήθηκαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μείωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ενδεχομένως και για κατάργηση των συνδικάτων. Βλέπουμε συνθήματα όπως ανταγωνιστικότητα οι μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά πρέπει να κάνουν απολύσεις. Κοιτάξτε, βαδίζει προς κατάργηση το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα και μας λένε ότι τα συνδικάτα δεν χρησιμεύουν πουθενά. Γιατί να ψηφίζει τότε ο Ευρωπαίος πολίτης σε ευρωεκλογές. Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη να ευχαριστήσω τους τρεις ε, προσκεκλημένους μας. Πρόκειται βεβαίως για εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα. Έχω διαβάσει αρκετά για αυτές τις υποθέσεις ε, και απομένουν ακόμη πολλά να διαβάσω. Η Κομισιόν στη δήλωσή της σήμερα είπε ότι ο κανονισμός, αν υπάρξει, θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα. Όμως Πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων για το ποια είναι τα προβλήματα. Μήπως λοιπόν μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ σας όσον αφορά το ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα για εμάνα. Δεύτερον, μας έχουν πει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει ιεράρχηση των δικαιωμάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης ε, και των δικαιωμάτων ελευθερίας ε, κίνησης. Όμως, από ό,τι φαίνεται με τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου, προτιμάει τις οικονομικές ελευθερίες και μας λέει ότι δεν είναι απόλυτο δικαίωμα το δικαίωμα της συλλογικής δράσης. Ρωτάω λοιπόν και εγώ μήπως το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών επίσης δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Επίσης, μας είπατε ότι άλλαξε η νομοθεσία στη Σουηδία. Αν υπάρξει άλλη μια υπόθεση Λαβάλ αύριο για τη Σουηδία, τι θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ κύριο Στέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές. Δεν έχω ερωτήσεις. Ε, προ την Business Europe και στην ε, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, γιατί οι θέσει του είναι ξεκάθαρε και είναι γραπτέ, αν θέλετε. Ε, έχω όμω ερωτήσει προ την Επιτροπή. Πρώτον, θα μπορούσαμε να έχουμε και γραπτά την προφορική ομιλία. Για να δούμε, μήπως αν κάτσουμε να διαβάσουμε με την ησυχία μας αυτή την ομιλία ε, και τουλάχιστον εγώ ξεκαθαρίζω τις αμφιβολίες μου όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής. Πάντως, σε ένα λεπτό, έτσι θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είναι θεμελιώδης. Άκουσα, αν κατάλαβα καλά από την, την ομιλία της Επιτροπής, ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν παραβίασαν οι αποφάσεις και δεν έχουν σε με κανένα ε, δικαίωμα ε, ε, των εργαζομένων. Αλλά κοιτάξτε, ακούγοντας τι λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, τι λένε τα συνδικάτα, ε, εδώ δεν πρόκειται μόνο πρόβλημα για τη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία, όπου παραβιάζονται τα κοινωνικά του δικαιώματα, ε, ιστορική παράδοση ε, των σωματείων, η δυνατότητα συλλογική δράση. Αλλά εδώ μιλάμε για συμβάσει πολύ σημαντικέ, όπω για παράδειγμα η σύμβαση του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασία υπαριθμών 87. Το λέει η ίδια η οργάνωση. Όπου εδώ ε, αναφέρεται το δικαίωμα τη απεργία. στοιχεία που έχουν να κάνουν επίση με την ελευθερία εγκατάσταση τα κτλ. Μα οι περιορισμοί στο δικαίωμα της απεργίας είναι πολύ ξεκάθαρες και, είναι πολύ ξεκάθαρες ε, και έχουν να κάνουν με οικονομικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση, αν θέλετε, ε, της, ε, ε, της αντίθεσης που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Και τα λέει αυτά η Παγκόσμια Οργάνωση της Εργασίας, δεν λέω εγώ. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Λέει ότι ε, δεν αποκλείεται η αναθεώρηση, αλλά η επιχειρηματολογία τη αποκλείει την αναθεώρηση. Είναι αλήθεια ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το μελετήσουμε με περισσότερη ησυχία. Ότι πρέπει να κάνουμε μια αυστηρή και επιστημονική προσέγγιση. Αλλά σα παρακαλώ, από τη μία, ε, όλα τα επιχειρήματα τη Επιτροπή να, είναι κατά τη αναθεώρηση και την άλλη να λέει ότι ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε την αναθεώρηση. Ε, όχι. Ε, το θέτει καθαρά ως πρόβλημα εφαρμογής. Όταν είναι προφανές ότι η οδηγία αυτή θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, στοιχειώδη θέματα του εργατικού δικαίου. Ε, έρχεται σε, σε, σε, τρομερό πρόβλημα με την ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τε, ε, εν πάση περιπτώσει πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά και υπάρχουν τρομερά προβλήματα στον αφορά την ερμηνεία τους. Άρα ε, δεν θέλουμε απλά και μόνο εφαρμοστικό κανονισμό. Θέλουμε κάτι περισσότερο. Θέλουμε διασαφήνιση. Μα πώ θα γίνει η διασαφήνιση ε, τη ερμηνεία του δικαστηρίου, αν δεν αλλάξει ο κανόνα και η νομοθεσία που οδήγησε στην απόφαση του δικαστηρίου. Και πώ θα αποφύγουμε, κύριε Πρόεδρε. Μα λέτε ότι με την εθνική νομοθεσία ε, ξεκαθαρίστηκαν τα προβλήματα. Όχι, όχι, τα προβλήματα εξακολουθούν να προκύπτουν. Μα τώρα ε, έχουμε μία νέα υπόθεση, σαν το Σπαλότα και άλλοι. Θα, θα ακολουθήσουν και άλλε υποθέσει. Γιατί αυτή η οδηγία, κύριε Πρόεδρε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ε, ε, ε, χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα απλό εφαρμοστικό κανονισμό. Ε, Ο κ. Κοφεράτη, τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα αυτές τις τελευταίες ε, δύο ημέρες ε, ε, πολλούς επένους στο κείμενο του Μάριο Μόντε και στο, έγγραφο του, κυρίου, του Μάριο Μόντε για την Επιτροπή. Αν το πιο καινοτόμο τμήμα μπορούσε να εφαρμοστεί, τότε αναπόφευκτα θα, θα διηθούν συμπέρασμα ότι χρειάζεται όχι μόνο προσαρμογή οδηγία, αλλά ριζική αλλαγή. Γιατί κατά την άποψή μου δεν υπάρχει εσωτερική αγορά αν δεν υπάρχει ισορροπία που ζητάει και ο ίδιος ο Μόντι ανάμεσα στα οικονομικά δικαιώματα και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί χωρίς αυτή την ισορροπία είναι αναπόφευκτο το dumping. Επειδή η κινητικότητα ε, φέρνει σε αντιπαράθεση, αν θέλετε, μοντέλα κοινωνικής εκπροσώπησης, ε, ε, εκπροσώπησης συμφερόντων, ακόμα και εκτιμένα δικαιώματα στην καθημερινή πρακτική που ε, μέσα από τις, ε, ε, με, την πάροδο των χρόνων και την πάροδο των δεκαετιών διαμορφώθηκαν με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πλέον είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, αν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη συλλογική σύμβαση και διαπραγμάτευση, ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα στην απεργία και ε, το συναφές δικαίωμα που έχει να κάνει με την εκπροσώπηση. Γιατί η συλλογική διαπραγματεύση, το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί. Από ποιον. Ποιος ε, έχει το, ε, αυτός που δέχεται το αποτέλεσμα είναι ο εργαζόμενος αλλά κοιτάξτε εδώ μιλάμε για ισομερή εκπροσώπηση εργαζόμενη και επιχείρηση και εδώ είναι φυσιολογικό όταν μιλάμε για τη διαπραγμάτευση να μιλάμε και για συγκρούσεις και εδώ βασικό εργαλείο είναι η υπεργία άρα αν δεν ε, συνδεθούν διαφορετικά αυτές οι πτυχές, θα καταλήξουμε στο να υποστηρίζουμε μόνο την εσωτερική αγορά και την επαναπρόθεσή της, χωρίς τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Εγώ θέλω να κάνω μια σύντομη ερώτηση για την ε, ε, εφαρμοστική οδηγία. Γιατί στην πρότασή σας σε τι αναφέραστε. Γιατί ε, είχα την εντύπωση ότι άμα δεν ξεκινήσουμε το ζήτημα τη συμμόρφωση και τη εφαρμογή, μπορεί να γίνει αναθεώρηση, εντάξει. Αλλά αν δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, τότε δεν ξέρουμε καν αν απαιτείται η αναθεώρηση. Μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερα. Ε, δύο λεπτά ε, ε έχουμε συνολικά, άρα ένα λεπτό ο καθένα για να συνοψίσει. Ξεκινάω με την ETUC. I will use my... Θα χρησιμοποιήσω το ένα λεπτό για να επιβεβαιώσω ότι τα ερωτήματα της κυρίας Χάρκιν είναι σωστά και πρέπει να απαντηθούν. Περιμένω πότε θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ναι, κανένα δικαίωμα δεν είναι απόλυτο, ενδεχομένως το δικαίωμα στη ζωή, αλλά ακόμη και αυτό το συζητάμε μερικές φορές. Όμως εδώ έχουμε μία ισορροπία. Μιλάει το δικαστήριο για ισορροπία, όλοι ζητάνε ισορροπία, αλλά εγώ δεν βλέπω ισορροπία εδώ. Βλέπουμε ότι οι οργανωμένοι εργαζόμενοι και όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους διασυνοριακά επειδή θέλουμε ισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες για να μην θυμώσουν με τους μετανάστες για παράδειγμα Θέλουμε να στηρίξουν και οι εργαζόμενοι τα ανοιχτά σύνορα και την εσωτερική αγορά, αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε δράση. Θα μου πείτε τι γίνεται με το δικαίωμα μιας χώρας να μετακινείται διασυνοριακά, να αλλάξει έδρα. Κανένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει προστασία της συνθήκης και δεν μπορούν να την επικαλούνται έναντι όλων που αντιτίθεται σε αυτούς. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιούν για να αποφύγουν τις συλλογικέ συμφωνίες, τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Αν ο μόνος λόγος που μετακινείστε που αλλάζετε έδρα είναι για να πληρώνετε χαμηλότερες μισθούς, τότε αυτό αντιβαίνει στο σκοπό της συνθήκης. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Χάρκιν για την ερώτηση που έθεσε. Ευχαριστώ. Κύριε Μαξίμ Τσερούτη, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Μου ζητήσατε να εντοπίσω τα προβλήματα. Δύο είναι τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και δικαίωμα συλλογική δράσης. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το δικαστήριο, όμως τα κριτήρια που χρησιμοποιεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτά που θέλετε. Υπάρχει το δικαίωμα δράσης των εργαζομένων. Θα πρέπει να δούμε τι ισορροπία θα πρέπει να επιτύχουμε. Μετά, πού εφαρμόζεται η οδηγία για τις αποσπάσεις. Για να υπάρξει ισορροπία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν ήταν σαφές αυτό γιατί δεν συμμετείχαν στις συλλογικέ συμβάσεις αυτής οι εταιρείες. Όμως αυτό το πρόβλημα τώρα δεν υπάρχει πλέον. Έγινε δηλαδή αυτό. Άλλο ερώτημα. Όταν υπάρχει συλλογική συμφωνία γενική, μπορεί αυτή να υπερβεί τους κανόνες που ισχύουν από την οδηγία. Νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά βεβαίως πάντα πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση με την οδηγία για τις αποσπάσεις. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και συζητήσει με την ΕΤΟΥΚ έχουν ήδη επιληθεί επαρκώς και γι' αυτό τώρα θέλουμε να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Business Europe, το πιο εύκολο ερώτημα είναι το αν θα σας διαθέσω το κείμενο της δήλωσής μου. Ναι, μπορώ να το κάνω. Τώρα, για τα υπόλοιπα πολλές παρεμβάσεις θεωρούν ότι η μισθή των αποσπασμένων εργαζομένων είναι πολύ χαμηλότερη από τον εντόπιων εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε αποδείξεις. Θέλουμε περισσότερες αποδείξεις για να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Επί της αρχής πάντως η οδηγία θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποφυγή τέτοιων καταστάσεων γιατί έχει συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για τον ελάχιστο μισθό, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για το χρόνο εργασίας κτλ. Και ο ελάχιστος μισθός πρέπει να ορίζεται είτε από την νομοθεσία είτε από Γενική Συλλογική Σύμβαση. Τι δεν κάνει η οδηγία. Δεν αντιτίθεται σε χρήση σε μη χρήση συλλογικών συμβάσεων που δεν εφαρμόζονται για το σύνολο της χώρας. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αν μια επιχείρηση πρέπει να πληρώνει υψηλότερους μισθούς στους αποσπασμένους εργαζόμενους, τότε αυτό θα δημιουργεί προβλήματα στους εργαζόμενους εντός της χώρας. Και βεβαίως αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των ε, εγχώριων επιχειρήσεων και των διασυνοριακών επιχειρήσεων. Κάτι που δεν θα το καταφέρναμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντως η εφαρμογή δεν είναι δύσκολη. Όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν γενικά, καλώς. Αν όμως δεν ισχύει αυτό, τότε υπερισχύει οδηγία. Όσον αφορά τώρα τον ILO, γνωρίζω την ε, γνώμη του ILO, που βεβαίως δεν είναι γνώμη του ILO αυτού καθ' αυτού, αλλά της ε, Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υπάρχει και αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην νομοθεσία για τις απεργίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για την οποία έχουν υπάρξει πολλές υποδείξεις αυτής της Επιτροπής στο παρελθόν. Όμως, όταν έχουμε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στη συνθήκη, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά δεν έχουμε παράγωγο δίκαιο που να καθορίζει πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται αυτές οι αρχές στην πράξη, δημιουργείται πρόβλημα, γιατί θέλουμε ισότιμη προστασία και των οικονομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς πρέπει να επιληθεί το θέμα με πρωτογενή νομοθεσία. Θα μπορούσε όμως η συνθήκη δεν δίνει αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετεί για το δικαίωμα απεργίας. Αυτό αναφέρεται σαφώς σε άρθρο της συνθήκης και γι' αυτό και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι σαφής στο πώς θα χειριστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εκεί είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητές μας και πρέπει να το λάβετε υπόψη. Παρόλα αυτά, οι συστάσεις της εκθέσεις ε, Μόντι πρέπει να εξεταστούν ενδελοχώς, το κάνουμε αυτό και σίγουρα δεν πρόκειται να αντισαγνοήσουμε όταν καταλήξουμε σε μια τελική λύση. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Μήπως μπορείτε να μας στείλετε την προφορική σας παρουσίαση και αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις από τους ε, ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να σας τις στείλουν γραπτός και να απαντήσετε κι εσείς γραπτός. Γιατί δυστυχώς ε, πρέπει να κλείσουμε εξαιτίας των μηνέων. Σας ευχαριστώ πάντως και τους τρεις για τις ε, παρουσιάσεις σας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ. Και η επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 23 Ιουνίου και Τρίτη 24. Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 3.